that uh, Geoffrey cannot wait for... Πάντα χαίρομαι που ο Τζέφρι δεν μπορεί να περιμένει με ανυπομονησία προσμένει τις περαιτέρω δράσεις της ε, εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λέει ο Πρόεδρος. Μάλιστα. Κυρίες και κύριοι, ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Και τώρα θα περάσουμε στο σημείο ganze Liter der Anträge brauche ich. Und ich brauche auch diese. Ja. Für die Delegation habe ich schon parat. Und ich brauche auch das, wo das, diese Anträge. Wir beginnen mit dem. Ξεκινάμε λοιπόν με την έκθεση για την Ιαπωνία. Προβλέπετε στην ημερήσια διάταξη στο σημείο 10. Εισηγητής, ο κύριος Πέτερλε. Θέλετε να πάρετε το λόγο? Ε, ε, Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένο που συμφωνήσαμε και συμφωνήσατε κι εσείς με τη γραμμή που αντικατοπτρίζεται και στον, στη λίστα ψηφοφορία. Πρέπει να πω ότι δεν θα συμφωνήσω με νέες τροπολογίες και σε ό,τι αφορά συγκεκριμένα τις παλακίδες είναι σαφές τι έκανε ο Πρωθυπουργός Άντε πρόσφατα με τη δήλωσή του για το θέμα αυτό. Δεν υπάρχει λόγος να σχολιάσουμε δικές του δηλώσεις. Θα έλεγα λοιπόν να ακολουθήσουμε τη γραμμή που συμφωνήθηκε και η έκθεση αυτή να προσανατολίζεται προς το μέλλον Α μην ασχοληθούμε με κρεμή ζητήματα του παρελθόντο. Αυτή είναι η γραμμή μου. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ πολύ. Να ξεκινήσουμε λοιπόν. Η 13, τροπολογία 13, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 14, υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 15 μαζί με την προφορική τροπολογία 3, υπέρ.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 Κατά αποχές εγκρίνεται. 31 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 32 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 33 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 34 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 35 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 36 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 38 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία 7 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 39 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 40 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 41 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 42 υπέρ. Και 30 μαζί. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 43 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 44 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται προφορική τροπολογία 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 45 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 46 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 3 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 4 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία 2 υπέρ. Κατά. Αποχέ εγκρίνεται 6 υπέρ. Κατά. Αποχέ εγκρίνεται 7 υπέρ. Κατά. Αποχέ απορρίπτεται 8 υπέρ. Κατά. Αποχέ εγκρίνεται 9 υπέρ. Κατά. Αποχέ εγκρίνεται 10 υπέρ. Κα... Α, καταπίπτει. Συμβαστική 1 υπέρ. Κατά. Αποχέ εγκρίνεται 1 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται, 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία για το σύνολο του κειμένου παρακαλώ. Έναρξη της ψηφοφορίας. Α, ναι, και η κάρτα μου λέει ο Πρόεδρος. Abstimmung ist geschlossen. Πέρα της 47 υπέρ, καμία ψήφο κατά και 9 αποχέ. Συγχαρητήρια λοιπόν στον εισηγητή. Και τώρα περνάμε στη συμφωνία πλαίσια μεταξύ τη Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Γεωργία. ηλεκτρονική ψηφοφορία παρακαλώ, έναρξη ψηφοφορία. ψηφοφορίας. Να προτείνω και να πω ότι αυτό το αποτέλεσμα είναι καλύτερο και από αυτό το δημοψήφισμα της Κρυμαίας. Ομόφωνα εγκρίνεται. Συγχαρητήρια. Συνάδελφε Λίζεκ. Και τώρα περνάμε στο σημείο 12 της ημερήσιας διάταξης η υπόθεση Μαγνίτσκι. Καμία παρατηρήση, σχόλιο της εισηγήτριας, όχι. Τροπολογία 1, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 2, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η 3 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Η 4 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 5 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 6 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 10 σε δύο τμήματα, πρώτο τμήμα υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Η 11 γλωσσολογικής φύσεως. Και τώρα περνάμε στη 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Και τώρα περνάμε στην 48. 49 διορθώνει. Πότο Σασιεβίτς. 49 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 50 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Και τώρα τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Παρακαλώ, έναρξη ψηφοφορίας. Καμίλε τι, Abstimmung ist ψηφοφορίας. 53 ψήφοι υπέρ, μία κατά, δύο αποχές, εγκρίνεται. Συγχαρητήρια, κυρία Γιουλάντ Και τώρα περνάμε στο 13 της της διάταξης σε ό,τι αφορά τα Ηνωμένα Έθνη και η συγκεκριτή είναι ο κ. Λάμπστορφ, δεν ξέρω, εδώ είναι. Όχι, κάποιον άλλον θα εκνευρίζει. Ποιος τον ε, εκπροσωπεί εδώ, η κυρία Νέιντς. ας υποθέσουμε ότι μας παρακολουθεί με το πνεύμα ο κύριος Λάμστατ. Και περνάμε στη συμβαστική α, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Και τώρα περνάμε στην 11, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 13, υπέρ. Θέλετε να ελέγξουμε την 11. Ω, όπως θέλετε. Έναρξη ψηφοφορία παρακαλώ ηλεκτρονική για την τροπολογία υπεριθμών 11. Πέρα. Ναι. Μα ποιο ζήτησε έλεγχο. Ποιο ζήτησε έλεγχο. Να δω. Εγκρίνεται 13 υπέρ κατά άποχες έλεγχος παρακαλώ γιατί δεν ψήφισαν οι σοσιαλιστές. Μαρίτσα, μου το υποσχεθήκατε. Αυτά που λέγαμε μεταξύ μας στην κρεβατοκάμαρα δεν πρέπει να τα αναβιάρουν προς τα έξω. Τα ενίκο μη ενδύμω. 36 ψήφοι υπέρ, 21 κατά. Ε, ε, είναι και το θέμα, ξέρετε, το άλλο να κάνεις μια υπόσχεση και άλλο να την τηρήσεις. Και έτσι περνάμε λοιπόν στην τροπολογία πράγμα 12 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική B υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 15 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική C, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 20. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 21. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 22. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 24. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 25. Υπέρ.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 Κατά αποχές εγκρίνεται. 34 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Σεμιβαστική ή e. υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 38 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 40, 39, συγγνώμη, υπέρ, κατά, αποχές, έγκρινεται, 40, υπέρ, κατά, αποχές, έγκρινεται, 41, υπέρ, κατά, αποχές, έγκρινεται, 42, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 43 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 44 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 45 υπέρ. Πρώτο τμήμα, συγγνώμη, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική F. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Και τώρα περνάμε στη συμβαστική G. Υπέρ.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 κατά αποχές εγκρίνεται. Και τώρα περνάμε στην τροπολογία 55 δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 57 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική I. Ι. Υπέρ. Αποχές εγκρίνεται. 59 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα παρακαλώ υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 61 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική J υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 64 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Διαδικαστικό, διαδικαστικό κύριε Πρόεδρο. No, we voted it. We voted it. We voted it. Yes. That we voted. And was yes. Ψηφίσαμε και ήταν υπέρ. Το αποτέλεσμα ήταν θετικό. Uh, we have to check now 64. 64. Την 64 θέλετε να ελέγξουμε. Ωραία. Yes, geschlossen. 35 υπέρ, 21 κατά, εγκρίνεται 65 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 66 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η φιλελεύθερη ψήφιση είναι υπέρ. Α, και είναι και όχι ψήφισαν.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 81 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 83 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 84 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 83 υπέρ κατά αποχές Νομίζω ότι εγκρίνεται, αλλά αν θέλετε το ελέγχουμε κιόλα. Ωραία. 4 υπέρ. Ναι, εγκρίθηκε, εγκρίθηκε λοιπόν. Η 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεβένα καλύπτεται. Δεβε 2 υπέρ. Όχι, τουλάχιστον δική μου η ομάδα έχει διαφορετική άποψη για διάφορες τροπολογίες. ΔΕΒΕ 2 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. ΔΕΒΕ 6 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. ΔΕΒΕ 8 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. ΔΕΒΕ 9 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. ΔΕΒΕ 11 υπέρ. Κατά. Οι φιλελεύθεροι το κόψα μου. Δεν ψηφίζουν. Δεν 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Έλεγχος. ΔΕΒ 11 παρακαλώ, ηλεκτρονικός έλεγχος. Die Abstimmung ist geschlossen. Πέρα της ψηφοφορίας. 36 υπέρ, 21 ψήφι κατά, εγκρίνεται. 12 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. ΔΕΒΕ 13 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, απορρίπτεται. ΔΕΒΕ 16 υπέρ. Κατά. Αποχές. ΔΕΒΕ 16 παρακαλώ υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται, εγκρίνεται. 17, υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Ας ελέγξουμε λοιπόν την ΤΕΒΕ 17. Πέρας. 21 ψηφί υπέρ, 36 κατά. Ντέβε 19 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Και τώρα περνάμε στην ΔΕΒΕ 21 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. ΔΕΒΕ 22 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Και τώρα περνάμε λοιπόν στην τελική ψηφοφορία έναξη της ψηφοφορίας. Και έτσι περνάμε στο 14 της ημερής της διάταξης. Πέρασε της ψηφοφορίας, αφού έχει φύγει ο κ. Λάμπσορφ, 46 ψήφοι υπέρ, 7 κάρτα, 2 απόχες, συγχαρητήρια. Και τώρα να περάσουμε στην... στο σύναψη πρωτοκόλλου της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ Ευρωπαϊκών Κοινωνιτήτων και της Δημοκρατίας του Μαυροβουνίου. ηλεκτρονική ψηφοφορία, παρακαλώ. Πέρας. Σαράντα εννέα ψήφι υπέρ, μηδέν αποχές, μηδέν ψήφι κατά. Συγχαρητήρια και στους Κροάτες φίλους μας. Και έτσι λοιπόν περνάμε στη 15, στο 15 της υπηρεσίας διάταξης. Ιράν. Σύσταση προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Τροπολογία 42 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 43 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος παρακαλώ. Πέρας ψηφοφορίες. Είκοσι έξι υπέρ, είκοσι έξι κατά, απορρίπτεται. 4 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 45 υπέρ. Σαράντα πέντε. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 46 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 47 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Μα έχει προσυπογράψει η πλειοψηφία της Επιτροπής. Τι είναι τώρα αυτό. Έλεγχος. Πέρας. Πέρας. Δίκιο είχατε. 26 υπέρ, 26 κατά. Απορρίπτεται.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 27 ψήφοι υπέρ, 25 κατά, εγκρίνεται. Η 49 ήταν αυτή. Η 50 υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. Έλεγχος ζητείται. Die Abstimmung ist Εγκρίνεται. Να συγχαρώ την Ιρανική αποστολή. Σε 52 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 53 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος παρακαλώ. auch mit 27 zu 26 angenommen. Das 27 υπέρ, 26 κατά εγκρίνεται επίσης. Συμβαστική 1. Υπέρ. Κατά. Ε, εγκρίνεται. 63. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Και τώρα περνάμε στην 73. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 74. Υπέρ. 74 dafür. υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. 75 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 76 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και τώρα περνάμε στην τροπολογία 78. Όχι, συγγνώμη, 87. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 89 υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 4 υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. 97 υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 5 υπέρ. Κατά, αποχές, Έλεγχος παρακαλώ, ηλεκτρονικός. Πέρας ψηφορίας. 26 υπέρ, 25 κατά εγκρίνεται. 107. Τι συμβιβασμοί είναι αυτοί που εγκρίνονται με μία ψήφο διαφορά μόνο. 107 υπέρ. Κατά. Άποχες απορρίπτεται. 109 υπέρ. Κατά. Αποχές ε, απορρίπτεται. 110 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 111 υπέρ. Κατά. Άποχες. Δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα. Πέρα ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 112 υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. Α, εγκρίνεται. Α, απορρίπτεται. Να το ελέγξουμε παρακαλώ. Να ελέγξουμε την 112. ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 113 υπέρ. Κατά. απόχέ απορρίπτεται. Συμβαστική 6 υπέρ. Κατά. απόχέ εγκρίνεται. 114. Όχι, όχι, όχι, όχι. 122 υπέρ. Κατά. απόχέ. 122, 122. χωρίς την προφορική τροπολογία. Την 122 ψηφίζουμε μόνο. Όπως έχει. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. 12 υπέρ 40 κατά απορρίπτεται. 124 υπέρ Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 9. Συμβαστική 9. Υπέρ. Κατά. Κύριε Κέλαμ. Uh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η τροπολογία 140 κατά τη γνώμη μου δεν καλύπτεται από τη συμβαστική τροπολογία 7, οπότε θα ήθελα να ψηφίσουμε ξεχωριστά την 140. Συγήτρια, έχει αμφιβολίες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η τροπολογία 140 καλύπτεται από τη συμβαστική τροπολογία. Κύριε Κέλλα, Η τροπολογία 140 δίνει κάποια ποσοτικά στοιχεία για τις εκτελέσεις, ε, κάποιους αριθμούς για τις εκτελέσεις στο Ιράν. Υπάρχουν όμως άλλα στοιχεία που δίνουν ε, άλλους αριθμούς. Απλώς η συμβαστική λύση μιλάει για μεγάλο, βαθμό, μεγάλο αριθμό εκτελέσεων. Δεν έχουμε αξιόπιστα ακριβή στοιχεία για τον ακριβή αριθμό εκτελέσεων. Προτιμώ να πούμε μεγάλος αριθμός, υψηλός αριθμός εκτελέσεων παρά να δεχτούμε την τροπολογία του κ. Κέλλαμ που δίνει συγκεκριμένο αριθμό που δεν είναι όμως εξακριβωμένος, γιατί άλλα στοιχεία είναι αντιφατικά. Με βάση τη, τον κατάλογο της α, γραμματείας, δεν φαίνεται να καλύπτει η τροπολογία 140 από την συμβαστική τροπολογία 7. Μπορεί να καταπίπτουμε με την έγκριση της συμβαστική τροπολογίας, αλλά από τη στιγμή που δεν καλύπτεται ρητά από τη συμβαστική τροπολογία 7 με βάση το κατάλογο ψηφοφορίας, θα ήθελα να την ψηφίσουμε ξεχωριστά την τροπολογία 140. Κυρία Μουνής. Έγινε λάθος στον κατάλογο της ψηφοφορίας. Δεν αναφέρθηκε το 140, τροπολογία 140. Το περιεχόμενο όμως της τροπολογίας 140 καλύπτεται από τη συμβαστική τροπολογία 7. Όντως, ξεχάσαμε να βάλουμε τον αριθμό 140 στις τροπολογίες που καλύπτονται. Αλλά το περιεχόμενο, παραλαμβάνω, καλύπτεται, γιατί η συμβαστική τροπολογία μιλά για μεγάλο αριθμό εκτελέσεων. Ενώ η τροπολογία 140 μιλά για 650 εκτελέσεις. Η 127 τροπολογία μιλάει για 675. Η 119 τροπολογία μιλάει για 500 εκτελέσεις. Δεν υπάρχουν εξακριβωμένα και ακριβή αξιόπιστα στοιχεία για τον αριθμό των εκτελέσεων στο Ιράν. Προτιμώ να μιλούμε γενικά για μεγάλο αριθμό εκτελέσεων. Τώρα για το τι δεν αναφέρεται στο κατάλογο ψηφοφορία η 140 είναι λάθο. Παραλήθηκε κατά λάθο ε, η τροπολογία 140. Κύριο Κέλαμ. Διαφωνώ με την εισηγήτρια. Γιατί το νόημα της τροπολογίας 140 είναι να κάνουμε έκκληση προς τις ελληνικές αρχές να λάβουν υπόψη αυτά τα νούμερα. Η αλήθεια είναι ότι συγκεκριμένος αριθμός εκτελέσεων έχει πραγματοποιηθεί και θα πρέπει να τις αναφέρουμε συγκεκριμένα. Επιμένω λοιπόν στην ψηφοφορία της τροπολογίας 140 ξεχωριστά. Υπάρχει μήπως η εξή ε, δυνατότητα. Υπάρχουν κάποιες επιπλέον πληροφορίες σας σε ό,τι αφορά τη διεθνή αμνηστία, τα Ηνωμένα Έθνη, ότι εκφράζουν ανησυχία, ε, όχι μόνο ανησυχία, αλλά alarm. Ε, θα μπορούσαμε για το ΕΛΚ να αποτεχτούμε να κάνουμε μία ξεχωριστή ψηφοφορία για την διαφορετική διατύπωση, για να πούμε expresses alarm, προκειμένου να ακολουθήσουμε την εισηγήτρια σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο και τα αριθμητικά στοιχεία που δεν θέλουν να δοθούν αλλά να ψηφίσουμε και το θέμα αυτό που μας απασχολεί. Νομίζω ότι είναι δίκαια λύση. κυρία Μουνίτ που είναι εισηγήτρια να πάρει πρώτη το λόγο. Ευχαριστώ και ευχαριστώ και για την πρότασή σας κύριε Πρόεδρε. Θα μπορούσαμε όντως ε, εκεί που λέμε να εξακολουθεί να εκφράζει τη σοβαρή της ανησυχία αυτό λέει η συμβαστική τροπολογία. Εντάξει, να πούμε, έχει θορυβηθεί η κρούη των κόδωνα του κινδύνου. Αλλά την ε, σοβαρή μας ανησυχία και προβληματισμό την αναφέρουμε ήδη στη συμβαστική τροπολογία. Να προτείνω, επειδή η τελευταία πρόταση δεν περιλαμβάνεται σε καμία περίπτωση το συμβιβασμό, θα αποφασίσω ότι αυτό το ζήτημα για το great numbers ή πώς αναφέρεται συγκεκριμένα, high number, high number, υψηλός αριθμός. Αυτό λοιπόν το ε, περιλαμβάνουμε. Και αφαιρούμε λοιπόν τον αριθμητικά στοιχεία του ΚΕΛΑΜ και ψηφίζουμε το υπόλοιπο, τις υπόλοιπες διαφορές ε, ε, με τον συμβασμό και θα κάνουμε γλωσσική προσαρμογή, εντάξει. Ποιος λοιπόν υπό την έννοια αυτή υποστηρίζει την ε, τροπολογία Κέλαμ και Σία. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Έλεγχος. Μα σε κάποιες περιπτώσεις θα έπρεπε να δείχνει και κάποια ότι ευγένεια η συγγήτρια και ο συγγητή. Α, συγγνώμη, έκανα λάθος, λέει ο πρόεδρος. Πέρα ψηφοφορία. Και εγκρίνεται. Χωρίς τα αριθμητικά στοιχεία. Συμβιβαστική 9 υπέρ κατά αποχές έκρινεται η 156 ε, υπέρ κατά αποχές η 145 είναι το ίδιο, η ίδια ιστορία δεν αποδέχεται το έλεγχο, ότι καλύπτεται Δεν καλύπτεται. Δεν καλύπτεται. Πρέπει να ψηφίσουμε την 145, λέει ο πρόεδρο. Κύριε Μνήχ. Δεν έχω πρόβλημα να ψηφίσουμε τα πάντα. Εκτός από τις συμβαστικές τροπολογίες που έχουμε συμφωνήσει μετά και τι άλλε πολιτικέ ομάδες. Αλλά ο κατάλογος ψηφοφορία που έχει εκπονήσει η γραμματεία αναφέρει εκπίπτει, καταπίπτει εφόσον εγκριθεί συμβαστική τροπολογία 9. Η συμβαστική τροπολογία 9 εγκρίθηκε, άρα θα πρέπει να καταπέσει. Τώρα μην λέμε ποιες τροπολογίες καλύπτονται από ποιες συμβαστικές τροπολογίες, τα είπαμε από πριν. Κοιτάξτε, πρόκειται για ένα κατάλογο που την προετοιμάζει, τον προετοιμάζει η γραμματεία, αλλά τελικά αποφασίζει ο πρόεδρος. Καλή τώρα να δώσει... Ε, απεριόριστη πρόσβαση στον απεσταλμένο στο Ιράν. Αυτό δεν καλύπτεται από το συμβασμό και δεν κατανοώ γιατί είμαστε κατά του δικαιώματος αυτού νου για τον ειδικό απεσταλμένο των Ηνωμένων Εθνών. Κύριε Σαλαφράγκα. Κύριε Πρόεδρε, η, η Γραμματεία έχει στείλει mail στι πολιτικέ ομάδε λέγοντα ότι δεν καλύπτεται αυτή η τροπολογία και ότι θα πρέπει να την ψηφίσουμε ξεχωριστά. Λίγη σοβαρότητα παρακαλώ στι αποφάσει και στις, στα μηνύματα που μα έχει στείλει η γραμματεία. Κατά λάθο δεν καλύπτεται από τη συμβαστική τροπολογία. Η εντολή τη γραμματεία είναι να ψηφίσουμε ξεχωριστά την τροπολογία αυτή, εφόσον δεν καλύπτεται από τη συμβαστική τροπολογία αναφέρεται στην έκθεση στην συμβιβαστική τροπολογία καλύπτει την Ευρωπαϊκή Ένωση να υποστηρίξει πλήρως το έργο του δικού απαστηλμένου των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα αυτά στο Ιράν. Αυτό δεν καλύπτει την τροπολογία του ΕΛΚ. Τόσο απλό είναι. Μπορούμε να το προσθέσουμε ως δεύτερο τμήμα της πρότασης. Την πρόταση του ΕΛΚ, αν σωστά καταλαβαίνω, είναι ότι καλύπτει την Ευρωπαϊκή Ένωση να υποστηρίξει τον ειδικό απεσταλμένο του ΟΗΕ και καλεί το Ιράν να δώσει θεώρηση πρόσβαση στον ειδικό απεσταλμένο του ΟΗΕ στο Ιράν. Άμεσα. Αυτή είναι η πρόταση του Έλκαν, σωστά καταλαβαίνω. Το αποδεχόμαστε αυτό. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ας ψηφίσουμε. 145 υπέρ. Κατά. Άποχες. Ούτως λοιπόν αποφασίστηκε 156 ε, υπέρ. Κατά. Άποχες. 156 λέω. Ηλεκτρονικός έλεγχος. 28 υπέρ, 27 κατά. Η 156 54 εγκρίθηκε. 157 υπέρ. Κατά αποχές. 157 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 158 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 159 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 162 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 10 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 169. Όχι. Ναι. Υπέρ. Όχι. Καλύπτεται και αυτή. 170. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 171. Υπέρ. Κατά εγκρίνεται. 172. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 173. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 175. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 176. Υπέρ. Κατά αποχές έλεγχος. Γιατί είναι 185 Έλεγχος. Έλεγχος. Πέρασε. «27 υπέρ, 29 κατά, απορρίπτεται». Και τώρα περνάμε στην 176 υπέρ. Κατά. Άποχες. Έλεγχος. Πέρας. 25 υπέρ, 30 κατά, απορρίπτεται 198. Α, 177 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Α, 178 υπέρ. Α, καταπίπτει. Μπέλντερ κατά Κρόνμπεργκ. 12 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 13 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 14 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 15 υπέρ. Κατά αποχές έλεγχος παρακαλώ. Πέρας. Τριάντα υπέρ, 26 κατά, εγκρίνεται. Η 15 εγκρίθηκε και τώρα ψηφίζουμε το δεύτερο τμήμα της 16 μόνο υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ο 18 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 19 υπέρ. Κατά αποχές Απορρίπτεται. 20. Να ψηφίσουμε. 20 υπέρ. Κατά. Έλεγχος. εγκρίνεται 29 υπέρ 26 κατά. 21. Α, δεν χρειάζεται να το ψηφίσουμε. 23 υπέρ. Κατά. Άποχες. Έλεγχος. Πέρας. 31 υπέρ, 25 κατά. Εγκρίνεται. Και τώρα περνάμε στην 27 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 28 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 29 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 30 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 31 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 32 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 33. 36 μάλλον, υπέρ. Κατά. Αποχές, εγκρι... ε, κατα... απορρίπτεται. Θέλετε έλεγχο, ζητάτε έλεγχο. Για την 36. Πέρας. 26 υπέρ, 31 κατά, απορρίπτεται. 37 Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 39 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 41 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 1. Έλεγχος. Για τη 41. Πέρας. 20 υπέρ, 36 κατά. Να παρακαλέσω τους σοσιαλιστές να... Είναι οι βουλευτές αυτοί που θα ζητούν έλεγχο και όχι οι βοηθοί τους. Ένα υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δύο υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 3 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 4 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τι έγινε με τη 2 και την 3? Α, εγκρίνονται. 7 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 8 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 9 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 11 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία τώρα. Πέρα ψηφοφορίας. Η έκθεση απορρίπτεται. 25 ψήφοι υπέρ, 30 κατά. Mr. Shaki. Η κυρία Σχάκε και ο κύριος Πρέντα. Ευχαριστώ. Ήθελα να επισημάνω ότι όταν ε, ξεκινήσαμε να κοιτάζουμε τις τροπολογίες και ε, καταρτήσαμε τον κατάλογο ψηφοφορία. Ε, πρέπει να πω ότι οι συνάδελφοι ξέρουν ότι η συνδυασία αυτή μεταδίδεται στο διαδίκτυο και πολλοί κόσμοι παρακολουθεί. Λοιπόν, εδώ κατά τη διαδικασία βρήκαμε το ΕΛΚ και οι φιλελεύθεροι να ψηφίσουν κατά. Γιατί, θα ήθελα κάποια εξήγηση. Το γεγονό ότι το σώμα αυτό δεν είναι σε θέση να καταλήξει σε ένα κοινό ψήφισμα για το πώ η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να προσεγγίσει το Ιράν, νομίζω ότι είναι κάτι που είναι αρνητικό για μα στην πολιτική μα θητεία. Οπωσδήποτε, έχουμε ασχοληθεί με ανθρώπινα δικαιώματα, με τον πόλεμο στη Συρία, όπου το Ιράν διδραματίζει το ρόλο του κακού. Έχουμε κάνει προτάσεις για το πώς μπορεί να, γίνει επικοδομητική, να γίνουν επικοδομητικά ανοίγματα προς το Ιράν πέραν των πυρηνικών. Δεν καταλαβαίνω γιατί το ΕΛΚ διαπραγματεύεται και μετά ψηφίζει κατά αυτόν τον τρόπο. Πραγματικά είμαι σε σύγχυση και θα ήθελα μια εξήγηση. Νομίζω ότι είναι πολύ κακό δείγμα και σε πολύ κακή χρονική συγκυρία. Δεν έχω ερω... απάντηση σε αυτή την ερώτηση, Έχω για άλλο λόγο ζήτησα να μιλήσω. Να σας δώσω λοιπόν ποια είναι η προσωπική μου άποψη και να σας παρουσιάσω γιατί καταψήφισα. Μεταξύ άλλων η τροπολογία Losing Ernst. Εξ όσων γνωρίζω το Ιράν δεν είναι στη Μέση Ανατολή. Αλλά το θέμα της ε, ε, ζώνης ελεύθερης από πυρηνικά και το να ε, το θέσουμε αυτό στη συνάρτηση με το Ιράν ως ρεσιμότητα δεν βοηθάει το Ιράν και την κατάσταση. Θα προβούμε σε ενέργειες που δεν έχουν να κάνουμε ε, με το Ιράν και λυπάμαι που ε, εγκρίθηκε αυτή η πρόταση, αυτή η τροπολογία της ΓΚΟΕ από τους άλλους και γι' αυτό λοιπόν καταψήφισα την έκθεση. Και αυτό θα έπρεπε να το ξέρουμε, ότι πολλοί θα ψήφιζαν κατά της έκθεσης αν είχε γίνει μια προσπάθεια για ένα συμβασμό στο θέμα αυτό, θα, υπήρξε, θα υπήρχε άλλη στάση. Ήθελα όμως να έχω παρουσιάσω και τη δική μου άποψη. I δεν θα προσθέσω, Πρόεδρε, τη δική μου συμβόλαια στη συζήτηση αυτή, διότι ξανανοίγω ουσιαστικά το θέμα. Όμως, να πω ότι το ΕΛΚ και άλλες ομάδες της Επιτροπής, ίσως να συμφωνώ ότι αφού δεν συμφωνήσαμε σε κείμενο σήμερα, ίσως οι η συγγήτρια και οι σκιώδες μπορούν να συναντηθούν για να επεξεργαστούν περαιτέρω συμβαστικέ λύσεις. Εάν το κείμενο αυτό είναι μη παραδεκτό, θα μπορούσε να αναπευθεί. Γι' αυτό λοιπόν θα συνασπιστώ με τα σχόλια τη κυρία Χάκε. Έχει δίκιο ότι είναι πολύ κακή η εικόνα που δίνουμε αν δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε για το Ιράν και να συντονίσουμε τη δράση τη Ευρωπαϊκή Ένωση προ αυτή τη χώρα. Ο κύριο Αλαφράνκα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι είναι ατυχές που δεν καταλήξαμε σε συνένεση μεταξύ των πολιτικών ομάδων παρόλο που οι διαπραγματευτέ μα έχουν κάνει ό,τι καλύτερο μπορούσαν, αλλά δυστυχώ δεν πείσαμε του ίδιου μα του γείτονε μεταξύ πολιτικών ομάδων. Πάντω και ο πρόεδρο εξέφρασε την προσωπική του άποψη, κατά τη δική μα άποψη. Το μήνυμα που αποστέλουμε μετά την ψηφοφορία αυτή το μήνυμα που θα αποστέλαμε αν υπερψηφίζονταν το κείμενο αυτό θα ήταν θετικό προς το κυβερνών ε, καθεστώς. Οπότε γι' αυτό καταψηφίσαμε. Πάντως θα μπορούσαμε να επιδιώξουμε μεγαλύτερη συνένεση στην Ολομέλεια. Είναι σημαντικό το θέμα αυτό και θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε σε επίπεδο συνολικότερο. Όμως σήμερα το πρωί ε, το κείμενο του ψηφίσματος ε, δεν ε, ακολουθούσε τις παραμέτρους που είχαμε καθορίσει εμείς ως σημαντικές, οπότε δεν μπορούμε και εμείς να υπερψηφίσουμε ένα κείμενο που δεν συνάδει με τις αρχές μας, τις αρχές που έχουμε ορίσει. Θέλαμε να έχουμε ένα κείμενο που θα έχει τη στήριξη όλων των ομάδων, αλλά κάτι τέτοιο δεν καταστεί δυνατό. δεν αντικατοπτρίζει το κείμενο αυτό τις θέσεις της πολιτικής μας ομάδας. Γι' αυτό δυστυχώ δεν μπορούσαμε να στηρίξουμε το κείμενο και αυτό είναι ένα από τα στοιχεία της δημοκρατίας που βίαπουν το σώμα αυτό. Καλό θα ήταν... Καλό θα ήταν να προσπαθήσουμε να πετύχουμε συνένεση και στήριξη στην Ολομέλεια. Ελπίζω ότι θα είναι δυνατό αυτό. Πάντως προς στιγμή δεν είναι δυνατό να ψηφίσουμε το κείμενο όπως έχει προταθεί. Eh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, είχαμε πολλές συνεδριάσεις των ε, σκιωδών εισηγητών και νομίζω ότι η όλη διαδικασία ε, ήταν άκρος δημοκρατική, ακόμη και αν κάποιος τους απογοήτευσε. Γιατί κάποιοι συνάδελφοι δεν φαίνεται να συμμετείχαν ποτέ στις συναντήσεις αυτές. Ή τουλάχιστον δεν υπέβαλαν εγκαίρως στις τροπολογίες τους. Σε κάθε περίπτωση να αποστείλω ένα μήνυμα συνεργασίας για τα για το θέμα αυτό, όχι για το Ιράν, αλλά για τις σχέσεις και τη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Ιράν. Ένα θετικό μήνυμα ως προς τον μετριοπαθή ε, πρόεδρο και τη Συμφωνία της Γενέβης για το θέμα αυτό. Για το επίμαχο πυρηνικό πρόγραμμα. Τώρα, η έκθεση στηρίζεται σε τρεις άξονες. Καταρχήν υποστηρίζουμε την Συμφωνία για τα Πυρηνικά της Γενέβης, ε, το θέμα της ανάμειξης του Ιράν στις περιφερειακές συγκρούσεις και φυσικά ασκούμε δρυμύτατη κριτική και εκφράζουμε την αντίθεσή μας ε, ως προς την κατάσταση που επισημαίνουμε και που εστερνίζεται γενικώ η Ευρωπαϊκή Ένωση και τη θηλητεύουμε την παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων εκ μέρους του Ιράν. Όπως είπαν η κυρία Σάκια και η κυρία Κρόμπερ, καταλήξαμε σε συμβεστικές ε, τροπολογίες με τις πολιτικές ομάδες. Ακόμη και το, με τον κύριο Ζαλεύσκη είχα τηλεφωνική συνομιλία από το Στρασβούργο για να ε, οριστικοποιήσουμε τις διατυπώσεις ε, και τις λεπτομέρειές τους. Εγώ ως εισηγήτρια προσπάθησα να καταλήξω συμβαστική λύση. Την ανησυχία του δεν την είχα ακούσει στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, αλλά μπορούμε να πάει στιγμή να επανέλθουμε στις διαπραγματεύσεις και να προσθέσουμε πράγματα που δεν είχαν αναφερθεί τότε. Ευχαριστώ. Έχουν ζητήσει διάφοροι συνάδελφοι το λόγο, αλλά έχει καταφτάσει ήδη ο προσκεκλημένος μας. Αν είναι άποψη ολονών των εισηγητών και των συντονιστών, θα μπορούσα να διαπιστώσω ότι δεν ε, έγινε τελική ψηφοφορία. Και στην περίπτωση αυτή θα μπορούσαν οι ομάδες στο μεσημερινό διάλειμμα να συζητήσουν και να ψηφίσουν. Αν θα μπορούσαν να υποστηριχθούν αυτές οι προτάσεις του ΕΛΚ και από τις άλλες ομάδες. Αν ε, δεν συμβεί αυτό, θεωρώ ότι έχει λήξει το περιστατικό. Όχι, ο κύριος Αλαφράγκα. Κύριε Πρόεδρε, εμείς ψηφίσαμε το κείμενο και το απορρίψαμε. Δεν μπορούμε να λέμε ότι δεν το ψηφίσαμε. Το μόνο που θα μπορούσα να πω εκ μέρους ομάδας και να προσφέρω και θα ακούσουμε και τις άλλες πολιτικές ομάδες είναι να προσπαθήσουμε να καταλήξουμε συμφωνία και αν τα καταφέρουμε, αν καταφέρουμε να συμφωνήσουμε όλες οι πολιτικές ομάδες, τότε θα κάνουμε σαν να μην ψηφίσαμε και θα υποβάλουμε το κείμενο στην Ολομέλεια. Αν, εφόσον καταλήξουμε συμφωνία. Αλλά θα πρέπει να είναι ευρεία συμφωνία. Αλλιώ θα πρέπει να δεχτούμε το αποτέλεσμα τη ψηφοφορία, αν δεν καταφέρουμε να καταλήξουμε στη συμφωνία. Εγώ είμαι πρόθυμο να εργαστώ για να καταλήξουμε συμβαστική λύση. Αν όμω δεν καταφέρουμε να συμφωνήσουμε όλε οι πολιτικέ ομάδε, θα πρέπει να σεβαστούμε το αποτέλεσμα αυτή τη ψηφοφορία. θα προσπαθήσουμε να καταλήξουμε συμφωνία ενόψη τη Ολομέλεια, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε σαν να μην συνέβη τίποτα και να πάμε στην Ολομέλεια σαν να μην έχουμε ψηφίσει. Δεν μπορούμε να παραβλέπουμε το αποτέλεσμα τη ψηφοφορία, αλλά επαναλαμβάνω, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να καταλήξουμε στη συμφωνία πριν από την Ολομέλεια. Αν τα καταφέρουμε και συμφωνήσουμε όλε οι πολιτικέ ομάδε, καλώ. Έτσι θα ξεπεράσουμε το αδιέξοδο. Αν όμω δεν συμφωνήσουμε οι πολιτικέ ομάδε, θα πρέπει να σεβαστούμε το αποτέλεσμα τη ψηφοφορία. Αν λοιπόν σας ερμηνεύω σωστά, θα ήθελα να προτείνω το εξής. Θα γίνει μια απόπειρα συμφωνίας μεταξύ των πολιτικών ομάδων και αν καταλήξουμε συνενετικό κείμενο θα το ψηφίσουμε στις 31 Μαρτίου. Αν δεν τελεσφορήσουν οι συνομιλίες και δεν καταλήξουμε στη συμφωνία, δεν ε, θα υποβάλουμε κοινέ τροπολογίες. Αυτά λοιπόν να συμφωνείτε. Αλλά θα πρέπει οι πολιτικές ομάδες να προσπαθήσουν να τα βρουν, να συνεννοηθούν. Δεν μπορούμε να προβλέψουμε ψηφοφορία στη μήνυ ολομέλεια δεν έχουμε αρκετό χρόνο, θα πρέπει να περάσει τη δεύτερη ολομέλεια του Απρίλιο. Αλλά αυτό προϋποθέτει προσπάθεια συνεννόησης και διαλλακτικό πνεύμα για να καταλήξουμε σε ένα συνενετικό κείμενο και να μπορέσουμε να το υποβάλουμε στην Ολομέλεια με θετική σύσταση. Αυτά. Ευχαριστώ κύριο Σάριος Βόλσκι. Η Δούμα, ε, το Ρωσικό Κοινοβούλιο δηλαδή, υπερψήφισε την προσάρτηση της Κρυμαίας και μάλιστα ζήτησε ε, από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένες Πολιτείες να βάλουν όλα τα μέλη της Δούμα στο κατάλογο με τις κυρώσεις. Μάλιστα, θα ακολουθήσουμε τις, ε, τη συμβουλή αυτή. Πολύ αρνητικό μαντάτο και άλλη είδηση. Ο ρωσικός τύπος ανήγγειλε ότι ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου της Υπερδνηστερίας ζήτησε την προσάρτηση και αυτής της περιοχής στη Ρωσική Ομοσπονδία. Αυτά αναφέρει ο ρωσικός τύπος σήμερα. Δεύτερη λοιπόν δυσάρεστη είδηση για σήμερα. Η παράνομη προσάρτηση ε, χρειάζεται για να πραγματοποιηθεί, να οριστικοποιηθεί δύο με τρεις μήνες, έστω και εκ μέρους της Ρωσίας. Οπότε έχουμε καθήκον στο διάστημα αυτό να επιχειρήσουμε μια διπλωματική επίλυση της κρίσης. Okay, then let's wage war. Ας αλλάξουμε τότε... Ας αλλάξουμε... Κάποιο... Ας αλλάξουμε πόλεμο. Διότι σε αυτή την περίπτωση η Βρετανία θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει τη δυνατότητα υπογραφής μνημονίου. Κάτι που δεν θα ήταν εγγύηση. Kolleginnen und Kollegen, ich Συνάδελφοι, καλώς ορίζω τον κύριο Αχμαντ Αλγάρμπα, πρόεδρο του Εθνικού Συνασπισμού Συριακών Πανεστατικών και Αντιπολιστικών Δυνάμεων, σχετικά με την τρίτη επέτειο της έναρξης της Συριακής Επανάστασης, την οποία οι αντιπολιτικές δυνάμεις διεξάγουν με ειρηνικό τρόπο. Κύριε Αλγκάμπα, η ε, σύραξη στη Συρία δεν έχει σύγκριση με αυτό που έχουμε εμεί στην πρόσφατη ιστορία. Θα ήθελα να εκμεταλλευτούμε την ευκαιρία τη σημερινή σα προσέλευσης για το μπορεί να κάνει η διεθνή κοινότητα και να διευκολύνει την πολιτική επίλυση του θέματο σε μια σύγκρουση που ε, θα πρέπει να οδηγήσει σε μια δημοκρατική μετάβαση αυτή στη χώρα. Η κατάσταση αλλάζει διαρκώ και οι δυνατότητε εξέβρεση πολιτική λύση φαίνονται ισχνέ. Ωστόσο, η, η Γενέβη 2 και 1 και 2 απέτυχαν ω τώρα ω συνομιλίε. Η αντιπολίτευση έχει αποδυναμωθεί από στοιχεία ε, παραστατικά και από το καθεστώς και δεν υπάρχει και ενότητα στην, ε, στον αγώνα της. Ε, το, το καθεστώς μιλάει για, εθνικές, για εκλογές και δεν είναι σαφές ότι ο Ασάντ θα είναι υποψήφιος. Επίσης, το Κοινοβούλιο θα επιτρέψει την ε, υποβολή υποψηφιότητων από προεδρικούς υποψηφίους και δεν ξέρουμε ποια θα είναι, η εκβάση των εκλογών. Δεν ξέρουμε κατά πόσον το υπάρχον καθεστώ μπορεί να επιτρέψει την δημοκρατική μετάβαση τη χώρα. Οι δυνάμει τη αντιπολίτευση έχουν ε, δηλώσει ότι θα είναι ορόσημο το να γίνουν εθνικέ εκλογέ. Το τι μπορεί να γίνει για να αρχίσει η διαδικασία διαπραγμάτευση είναι κάτι πολύ σημαντικό και ποιε είναι οι δικέ σα απόψει για τι ε, προσπάθειε του ΙΕ να πιέσουν το καθεστώ του Ασάντ να επιστρέψουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων στη Γενέβη. Κύριε Αργκάρμπα, έχετε το λόγο. Καλημέρα σας. Καταρχά να ευχαριστήσω τους ε, διοργανωτές αυτής της συνάντησης. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση σε αυτή τη συνεδρίαση για να μπορέσουμε να συζητήσουμε για την επανάσταση στη Συρία. Σήμερα, στις 18 Μαρτίου μάλλον συγκεκριμένα του 2011, κλείνουμε τριετία από την έναρξη των θρηπαξιών τότε ξεκίνησε στην, Τέρα, στην Τέρα ε, η Επανάσταση όταν ε, βγήκαν στο δρόμο οι πολίτες και όλα ξεκίνησαν με παιδιά που έκαναν γραφίτες στους τοίχους των σχολείων τους. Τους τα συνέλαβαν, τους έβγαλαν τα νύχια για τιμωρία και έτσι ξεκίνησε η Επανάσταση στη Συρία και έχει κρατήσει μία ολόκληρη τριετία. οπωσδήποτε θα γνωρίζετε την έκταση που έχει πάρει η καταστροφική αυτή σύγκρουση και η ανθρωπιστική αυτή τραγωδία. Το κυβερνών καθεστώς εκτοξεύει πυράβλους ε, βαρέλια τα οποία έχουν μετατραπεί σε βόμβες, σε υλικό που εκτοξεύουν ε, αεροσκάφη. Στη Γενέβη προσήλθαμε με θετικό πνεύμα προκειμένου να εξέρουν μια πολιτική λύση και να μας επιτρέψει να ε, μεταβούμε σε μια περίοδο για να αλλάξει η σημερινή κατάσταση. Ο κύριος Ασάντ όμως δεν θέλει να γίνει μέρος της επίλυσης. Και αυτό που είδαμε στην πραγματικότητα να συμβαίνει όταν πήγαμε στη Γενέβη είναι πέραν των όσων προβλέπονταν. Δολοφονήθηκαν 5.000 άμαχοι, 5.000 πολίτες. Είναι αδιανόητο να διοργανωθούν διαπραγματεύσεις, ενώ γινόμαστε μάρτυρες μιας τέτοιας ε, συστηματικής σφαγίασης των πολιτών της χώρας. Και στην Γενέβη προσήλθαμε μετά από μια συνεδρία που διοργανώσαμε στο Παρίσι. Δεχτήκαμε να πάμε στην Γενέβη, αλλά εάν το καθεστώς οδηγήσει τις διαπραγματεύσεις σε αποτυχία, σε αυτή την περίπτωση, οι φίλοι και σύμμαχοί μας μεταξύ των οποίων η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη της, που είναι μέλη του βασικού, της βασικής ομάδας νερομοτεύσεων, θα πρέπει και οι φίλοι και οι μας να τοποθετηθούν, προκειμένου να <clears throat> υπερασπιστούν τους πολίτες και να τους προσφέρουν την στρατιωτική, ανθρωπιστική βοήθεια που τους χρειάζεται. Ο κύριος Λακτάρ Μπραήμι, ο ειδικό απεσταλμένος του ΟΗΕ για τη Συρία, έχει υποβάλει την έκθεσή του προτριημέρου και στην έκθεση όπως δημοσιεύτηκε αναφέρεται ότι το καθεστώς Αλασάντ θα πρέπει να θεωρηθεί υπεύθυνο για την αποτυχία των διαπραγματεύσεων. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, ο κ. Μπανκιμούν, επίσης ανέφερε και δήλωσε ότι η υποψηφιότητα του Μπασάρα Λασάντ για μια νέα θητεία θα αποτελούσε ισοπαίδωση κάθε δυνατότητας εξέβρεσης πολιτικής λύσης. Σήμερα έχουμε έρθει στο Ευρωκοινοβούλιο, έχουμε έρθει σε εσά για να σας γνωστοποιήσουμε όλες αυτές τις πληροφορίες, όλες αυτές τις λεπτομέρειες. Ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να μας στηρίξει με αντιπυραυλικό εξοπλισμό προκειμένου να μπορέσουμε να προστατέψουμε τον πληθυσμό της χώρας μας. Είστε κι εσείς μάρτυρες των όσων συμβαίνουν στο Χαλέπι. Μιλάμε για βόμβες, πραγματικές βόμβες που καταστρέφουν διαμερίσματα σε απλές πολυκατοικίες. Μιλάμε για πολίτες που χάνουν τη ζωή τους, για παιδιά που δολοφονούνται, γυναίκες ή επιζώντες που μένουν μέσα στα συντρίμια. Πρέπει να μπορέσουμε να υπερασπιστούμε το λαό μας, γι' αυτό χρειαζόμαστε τέτοιου είδους ε, στήριξη. Το ίδιο και η στρατιωτική αεροπορία που καθημερινά δολοφονεί τους ανθρώπους μας. Εσείς είστε και εσείς μάρτυρες της ε, ανθρωπιστικής αυτής τραγωδίας ε, στο, στη Συρία με 200.000 νεκρούς. Οι φορείς του ΙΕ αναγνωρίζουν ότι ο αριθμός των εσωτερικών μετατοπισμένων, εκτοπισμένων μάλλον, και των προσφύγων φτάνει τα 9 εκατομμύρια Σύρων. Το 1 τρίτο της επικράτειας της Συρίας έχει ισοπεδωθεί, είτε ε, ε, ολοσχερός είτε εν μέρη. Ερχόμαστε λοιπόν αντιμέτωποι με πραγματικές δυσκολίες. Δεν μπορούμε να προσφέρουμε αγωγή στους ε, τραυματισμένους, στους τραυματίες. Υπάρχουν κάποιοι σήμερα που έχουν μείνει, πολλοί που έχουν μείνει ανάπηροι από τις επιθέσεις. Γι' αυτό και εμείς έχουμε καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να προσφέρουμε κάποια, κάποιο είδους ε, υγειονομική περίθαλψη στους τραυματίες και τους ε, ακροτηριασμένους πολίτες. Κινούμαστε δυναμικά στο εσωτερικό της χώρας και κινητοποιούμε όλους τους πόρους που διαθέτουμε για να προσφέρουμε τις στοιχειώδεις αυτές υπηρεσίες του σύρους εντός της χώρας. Παρόλα αυτά, η τραγωδία έχει πάρει τέτοιες διαστάσεις που το σύνολο του δυναμικού μας και των πόρων μας δεν υπάρχει περίπτωση να αρκέσουν. Ακόμη και η ανθρωπιστική διάσταση. Γνωρίζετε σήμερα ότι ολόκληρες περιοχές της Συρίας βρίσκονται σε πολιορκία δεν υπάρχουν τρόφιμα, δεν υπάρχει πόσιμο νερό και δεν υπάρχουν φάρμακα σε αυτές τις περιοχές. Στη Συρία όσοι δεν έχουν δολοφονηθεί με τα όπλα δολοφονούνται μέσω της πείνας. σβήνουν σιγά σιγά λόγω του λοιμού. Ο Μπασάρα Λασάντ έχει ψηφίσει ουσιαστικά έναν, έχει εγκρίνει ένα δικό του νόμο. Ή θάνατος με τα όπλα ή θάνατος με την πείνα η παράδοση. Ποιο είναι το... ποια είναι πια η, το όραμά του για τον 21ο αιώνα. Να μας ε, σκοτώσει για τρίτη φορά. Δεν μπορεί να αποσιοποιηθεί λοιπόν αυτό το έγκλημα του καθεστώτος κατά του ίδιου του, του λαού. Ε, είμαστε εδώ για να σας αναφέρουμε το, τις διαστάσεις που έχει πάρει η ανθρωπιστική αυτή τραγωδία, το πόσο ανάγκη έχουμε από βοήθεια και ζητούμε την ε, έγκριση ενός ψηφίσματος στο επίπεδο του ΟΗΕ βάσει του άρθρου 7 του οργανισμού ώστε να δημιουργηθούν ανθρωπιστικοί διάδρομοι βάσει του κεφαλαίου συγκεκριμένα 7. Θέλουμε να υπάρξουν δεσμευτικά μέτρα με την εφαρμογή του ε, άρθρου 7 ώστε όλες οι ένοπλες δυνάμεις, παραστατικές ή όχι, που βρίσκονται στη Συρία να εγκαταλείψουν την επικράτεια της χώρας. Το καθεστώς της Συρίας επιτρέπει να έρχονται μισθοφόροι στη χώρα. Τους καλεί, τους υποδέχεται, υποδέχεται τους μισθοφόρους της Χεσμολάχ, αυτούς που ήρθαν από το Ιράκ και από την Ιρανική Εθνοφυλακή. η μισθοφόροι της Αλκάιντα στην οργάνωση για το Ισλαμικό κράτος της Συρίας και της Μέσης Ανατολής είναι επίσης στη χώρα μας. Προσπαθούμε να καταπολεμήσουμε αυτήν την τρομοκρατική οργάνωση η οποία στηρίζεται διοικητικά από την εξουσία της χώρας. Οι δυνάμεις μας έχουν αγωνιστεί ε, επί τετράμινο κατά της ε, τρομοκρατικής αυτής οργάνωσης και μπορέσαμε να, να απελευθερώσουμε το το Χαλέπι και το, ε, το Ιντλίμπ. Έχουμε διεξαγάγει μάχες ε, κατά της τρομοκρατικής αυτής οργάνωσης που την καλύπτουν άλλοι όμως. Την καλύπτει το καθεστώς, το επίσημο καθεστώς της χώρας. Πολεμάμε λοιπόν την τρομοκρατία αυτής της οργάνωσης που είναι παραφιάδα της Αλκάιντα. Προσπαθούμε να καταπολεμήσουμε την τρομοκρατία του καθεστώτος Αλ ε, Ασάντ και την ε, τρομοκρατία των Ιρανικών, των Ιρακινών και των δυνάμεων της Χεσμολάχ. Πρόκειται για ένα πραγματικό πόλεμο με τρεις αντιπάλους και στα πλαίσια αυτού του αγώνα νομίζω ότι αξίζουμε να λάβουμε κάποια βοήθεια. Βοήθεια χωρίς όρους. Αδιαμφισβήτητη βοήθεια στρατιωτική και ανθρωπιστική. Ήρθαμε εδώ σήμερα λοιπόν για να σας εκθέσουμε τις ανάγκες μας και για να σας πούμε ότι επιθυμούμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να μείνει στο πλευρό μας σε αυτήν την κρίσιμη καμπή στα πλαίσια του εθνικού συριακού συνασπισμού, αυτό που επιδιώκουμε είναι να δημιουργήσουμε ένα ελεύθερο δημοκρατικό κράτος που να βασίζεται στην πολυφωνία και την πλειοψηφία και όχι να κυβερνάται από την μειοψηφία. Ας μείνω στην αντιπολίτευση. Η χώρα αυτή να έχει μία κυβέρνηση που να προστατεύει τις ε, γυναίκες, τις μειονότητες, ε, μια χώρα που να εγγυάται τις ελευθερίες των ε, σύρων γυναικών και ανδρών. Ευχαριστώ. Thank you very much, uh, Mr. Ευχαριστούμε κύριε Αλτζάμπρα. Ευχαριστούμε για τη δήλωση σε αυτή στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στους ε, συναδέλφους μας ε, για να γίνει συζήτηση. Ο κύριος Χόουιτ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να καλωσορίσω τον κύριο Αλτζάρμπα εκ μέρους της Επιτροπής. Ε, ισχυρό θα ήθελα να σας στείλω, να απευθύνω θερμότατο χαιρετισμό εκ μέρους όλων των πολιτικών ομάδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δεν ισχυρίζεται νομίζω κανένας μας ότι η ευρωπαϊκή παγκόσμια απόκριση στην κρίση στη Συρία ήταν επαρκής. Και ε, συμφωνούμε με την έκκλησή σας ε, γιατί ε, αντιλαμβανόμαστε την ανάγκη να ληφθεί δράση το συντομότερο δυνατόν. Έχω κάποιες ερωτήσεις. Καταρχήν, παρακολουθούμε το δεύτερο γύρο διαπραγματεύσεων της Γενέβης και ευελπιστούμε ότι θα τελεσφορήσουν. Είμαι από αυτούς που ενδιαφέρονται και παρακολουθούν εκ του σύνεγγης το θέμα. Εσείς πώς βλέπετε εκ των έσω αυτές τις συνομιλίες του δεύτερου γύρου της Γενέβης. Πιστεύετε ότι θα σημειωθεί μια ε, επιτυχία, μια θετική καμπή. Γιατί μέχρι στιγμής δεν τελεσφόρησαν ε, τα διπλωματικά διαβήματα. Είναι νομίζω σημαντικό να απαντηθούν αυτά τα ερωτήματα. Δεύτερη ερώτηση. Αφορά τη δική μας υποστήριξη εκ μέρου Ευρωπαϊκή Ένωση Ένωσης τη δική σα συμμαχία, στον Εθνικό Συνασπισμό δηλαδή των Επαναστατικών και Αντιπολιτευτικών Συριακών Δυνάμεων. Μία πιστεύω από τις δυσκολίε αυτής της διαδικασία χωρί να θέλω να σας ασκήσω προσωπική κριτική, ε, μία από τι δυσκολίε είναι η πολυμορφία της αντιπολίτευσης, η ανομοιογένεια που τη χαρακτηρίζει. Είναι ετερόκλητη και όχι ιδιαίτερα συντονισμένη αντιπολίτευση και ίσως δεν υπάρχει απαραίτητη ομαλότητα για να εξασφαλιστεί μια ε, σωστή μετάβαση. Δεν ξέρω αν θα το σχολιάζετε αυτό. Με ενδιαφέρουν πάντως ιδιαίτερα τα σχόλιά σου για το κατά πόσο η διπλωματία, η οικονομική στήριξη, η επιμελητιακή στήριξη που προσφέρουμε στον συνασπισμό της αντιπολίτευσής σας, αν είναι επαρκή αυτή η στήριξη. Γιατί ζητήσατε όπλα. Αυτό το ακούσαμε και δεν είναι ακόμη αυτή η δεδηλωμένη βούληση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να στείλει όπλα, αλλά ως προς τη στήριξη κάνουμε πολλά. Μπορούμε να κάνουμε περισσότερα κατά τη γνώμη σας. Δεν είναι επαρκή αυτή η στήριξη που έχουμε προσφέρει. Και θα μπορούσατε ειλικρινά να μας πείτε για τους τζιχαντιστές. Δηλαδή αυτούς που υποστηρίζουν την Αλκάιδα και που επίσης είναι κάπως συμπερδεμένοι στην αντιπολίτευση. Εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα είμαστε ευγνώμονες αν μας δίνετε μια έντιμη και ειλικρινή απάντηση, γιατί πολλά από τα κόμματα μας φοβούνται ότι μια ομάδα αχρίων και καταχραστών θα αντικατασταθούν από την άλλη. Αυτό φοβόμαστε. Ελπίζω να μεριμνήσετε να μην συμβεί κάτι τέτοιο. Και σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων θερμά για τις απαντήσεις που θα μας δώσετε και επίσης για όσα μας έχετε πει μέχρι στιγμής. Ευχαριστώ κύριε Χόουιτ. Η κυρία Σάκη έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι σημαντικό να συνεχίσουμε την αναζήτηση των λύσεων όσο δύσκολο και αν είναι κάτι τέτοιο και χαίρομαι για την ευκαιρία που είχαμε να ανταλλάξουμε απόψεις. Ποια είναι η γνώμη σας, τι πιθανότητες έχει η διαδικασία της Γενέβης να ευοδοθεί και ποιος θα είναι ο ρόλος σας σε αυτή τη διαδικασία. Επίσης, ποιος είναι ο ρόλος που κατά τη γνώμη σας θα διαδραματίσει το Ιράν. Γιατί μερικοί πιστεύουν ότι δεν νοείται λύση χωρίς την συμμετοχή της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν που ενεργά στηρίζει τους ε, μαχητές της Χεσμολάχ. Ε, και άλλοι πιστεύουν ότι η ανάμειξη του Ιράν θα περιπλέξει τα πράγματα. Εσείς τι πιστεύετε ότι είναι σωστό. Επίσης, ε, οι εξτρεμιστικές ε, τζιχαντιστικές ομάδες ε, μεγαλώνουν τη συμμετοχή τους, γιατί υπάρχει, υπάρχουν πληροφορίες για μεταξύ τους αντιπαράθεση. Τι θα γίνει στο έγκυς μέλλον. Γιατί δεν υπάρχει ένα ενιαίο μέτωπο τζιχαντιστών. Υπάρχουν μερικές εξτρεμιστικές ομάδες που είναι ακόμη πιο βίες και ριζοσπαστικές από άλλες. Και αυτό μας ανησυχεί ιδιαίτερος, γιατί θα αντιλαμβάνεστε ότι βρίσκονται σε διασταυρωμένα πειρά ε, οι κάτοικοι της Σύριας ε, μεταξύ ενός βίου και ε, εξτρεμιστικών ομάδων που δεν προσφέρουν μια πολύμορφη και δημοκρατική κοινωνία ως εναλλακτική λύση. Αυτό μας προβληματίζει ιδιαίτερος. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν από τους βασικούς συνεισφορείς των ανθρωπιστικών προγραμμάτων και της ανθρωπιστικής βοήθειας Φυσικά λυπούμαστε λοιπόν, ειλικρινά για το μεγάλο αριθμό των σύρων που εξαρτούνται από την ανθρωπιστική αυτή βοήθεια. Υπάρχουν, υπάρχει περιορισμό όμω στην πρόσβαση αυτή τη ανθρωπιστική βοήθεια. Εσεί ω δυνάμει αντιπολίτευση, πώ μπορείτε να εξασφαλίσετε απρόσκοπτη μετάβαση τη ανθρωπιστική βοήθεια σε περιοχέ που αυτή τη στιγμή είναι αποκλεισμένε και απομονωμένε. Αυτά είναι τα πιο σημαντικά θέματα. Επίσης συμμετοχή της ε, Τουρκίας, ε, της Ιορδανίας, του Λιβάνου, συμμετοχή των γειτονικών χωρών, ε, γιατί είναι σημαντική και αυτή η συμμετοχή, η συνεισφορά τους και η συμβολή τους στην καλύτερη δρομολόγηση των ανθρωπιστικών προγραμμάτων και της βοήθειας. Θα πρέπει να αλλάξουμε την, τον προσανατολισμό μας, αν κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο. Κύριος Άτκινς. Πρόεδρε, Ευχαριστώ πολύ να καλωσορίσω και εγώ τον κύριο Αλνταρμπά για την, ε, κατά την επίσκεψή του αυτή. Έχουμε μια έκφραση τα αγγλικά. Όταν υπάρχουν ε, πολλές πολιτικές αποκλήσεις, λέμε ότι καλό είναι να πηγαίνουμε με τα, δύο πόδια, με τα πόδια σε δύο βάρκες. Εδώ Υπάρχουν λοιπόν ανησυχίες από τους φυσικούς συμμάχους σας για το πόσο ανάμεικτα είναι τα προθέσεις και τα σχέδια στην ίδια την αντιπολίτευση πέραν του ίδιου του Αλασάντ. Εκτιμώ λοιπόν αυτό που, λέγεται, που, λέγεται, που λέτε ότι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η διάσπαση από της αντιπολίτευσης και να το καταγράψουμε. Το θέμα είναι όμως και η δράση της Ρωσίας στην περίπτωση της Συρίας που δεν θέλει να υπάρχει καμία παρέμβαση παρέμβαση. Ακριβώς αυτό που συμβαίνει κατά τα άλλα αυτή τη στιγμή. Αλλά είναι ενδιαφέρον και το ακούσαμε και σήμερα το πρωί από κάποιον. Είπατε κι εσείς ότι πρέπει να σημειωθεί, πρέπει να σημειωθεί η θέση της Κίνας ε, σε σχέση με την Ουκρανία. Δεδομένων των προβλημάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας στη Συρία με την ε, Ρωσία και την Κίνα, έχετε σκεφτεί εμέσως ή άμεσα με τη βοήθεια ενδεχομένως άλλων να κάνετε ανοίγματα προς την Κίνα. Πιστεύετε ότι θα μπορούσε αυτό να λειτουργήσει, θα σας έκλειναν την πόρτα στα μούτρα. Διότι εάν ξεπεράσετε αυτό το αδιέξοδο, αυτή τη συμφόρυνση που έχει, συμφόρυνση που έχει δημιουργηθεί στις διαπραγματεύσεις, πρέπει να αναζητήσετε ένα διαφορετικό τρόπο να προχωρήσετε και να ρωτιέμαι αν η Κίνα ήταν ενδεχομένως μια σωστή επιλογή. Ευχαριστώ πολύ κύριε Άτκινς. Σας ευχαριστώ κύριε Αλτζάμπα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που βρίσκεστε εδώ και είναι πάρα πολύ εντυπωσιακά αυτά που αναγκαστικά μας αναφέρατε και μας παρουσιάσατε. Εγώ προσωπικά θα ήθελα να πω πέρα κάθε αμφιβολία ότι το καθεστώς Ασάτ επεβίωση και θα πρέπει να εξαφανιστεί η δεν μπορεί να υπάρξει ειρήνη για τον λαό της Συρίας αλλά ένας Ρώσος συγγραφέα είχε πει κάποτε ότι όταν κάποιος φεύγει από ένα μνημείο, δεν ξέρουμε ποιος θα είναι ο επόμενος στο μνημείο αυτό. Και ίσως το επόμενο πρόσωπο να είναι ακόμα χειρότερο. Ό,τι θέλουμε μπορούμε να λέμε κατά του Ασάντ, αλλά τι έκανε το καθεστώς του, οι χριστιανοί ήταν κάπως ελεύθεροι και ζούσαν ελεύθεροι, ασκούσαν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα ελεύθεροι. Στη Δεμασκό είδα σε μια εκκλησία έναν ε, σταυρό φωτισμένο. Αυτό δεν το βλέπει κανείς εύκολα σε πολλές αραβικές χώρες. Γι' αυτό λοιπόν ρωτώ. Τι γίνεται σήμερα με τις θρησκευτικέ μειονότητες, με τους χριστιανούς στη Συρία και πώς πρόκειται να αντιμετωπιστούν εάν εσείς κερδίσετε το οποίο ασφαλώς σας το εύχομαι, αλλά απεύχομαι να κερδίσουν φονταμεταλλιστές οι οποίοι θα δολοφονήσουν τους χριστιανούς. Πώς εκτιμάτε λοιπόν το θέμα αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πέτερινγκ. Ο κύριος Σέβεριν έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και ευχαριστούμε και τον ε, κύριο Αλτζάρμπα για την παρουσίασή του, την ομιλία του την οποία παρακολούθησα με ιδιαίτερη προσοχή. Αν κατάλαβα καλά, πιστεύετε ότι η τελική λύση θα δοθεί με πολιτικό τρόπο και όχι με στρατιωτικό, ότι δεν νοείται στρατιωτική λύση εδώ. Σας κατάλαβα καλά ή μήπως έκανα μια παρεξήγηση, μια παρερμηνία. Πιστεύετε ότι ε, νοείται και στρατιωτική λύση για το διέξοδο ή μόνο πολιτική. Αν λοιπόν μια διέξοδος θα προέλθει μόνο από την ε, πολιτική λύση, θα ήθελα να μου το επιβεβαιώσετε. Και αν συμφωνείτε ότι μόνο πολιτική λύση νοείται ως εναλλακτική, τι είδους πολιτική λύση θεωρείτε ως εφικτή και βιώσιμη. Γιατί μας ενδιαφέρει πολύ η εκτίμησή σας ε, για το σημείο αυτό. Και επίσης, ποια είναι κατά τη γνώμη σας ακόμη τα προσκόμματα που εμπόδισαν την πρόοδο της ε, διαδικασίας της Γενέβης προς μια πολιτική λύση που θεωρείται ότι είναι σκόπιμη. Ευχαριστώ. Ο κύριος Λαντσμπέργκης, ο τελευταίος ομίλητης. I would like, Να σας ευχαριστήσω για τις πληροφορίες που μας δώσατε και για την ανταλλαγή αυτή απόψεων. Ήθελα να μου πείτε, τώρα υπάρχει κάποια πρόοδος σε σχέση με το θέμα των εγκλημάτων του ΑΣΑΤ κατά της ανθρωπότητας. Τα χημικά όπλα που χρησιμοποιήθηκαν κατά των πολιτών που αντιμάχονταν το καθεστώς. Τόσοι άνθρωποι, τόσα παιδιά έχασαν τη ζωή τους. για το διεθνές δικαστήριο. Υπάρχει, υπάρχει τέτοιο δικαστήριο για να εκδικαστεί η υπόθεση. Εάν ε, υπήρξε μπλοκάρισμα στο Συμβούλιο Ασφαλείας ή αλλού, τουλάχιστον η αντιπολίτευση στη Συρία δεν μπορεί να το παραβλέψει θα πρέπει να πιέσει τα δημοκρατικά καθεστώτα, να μην το επιτρέπουν αυτό. Καταλαβαίνετε, η Ρωσία συγκαλύπτει τέτοια εγκληματικά, τέτοιες εγκληματικές ενέργειες του καθεστώτος ε, του Αλασάντ. Ε, είναι τόσο παρετημένη και τόσο αναγκασμένη να ζει στο δικό της ολοκληρωτισμό που το θέμα αυτό θα έπρεπε να έχει τεθεί επιτάπητος εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Τέτοιο πράγμα είναι. Χημικά όπλα κατά των πολιτών και των παιδιών. Πού ε, έχει πάει η υπόθεση αυτή. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Λαντσμπαργκής. Κύριε Αλζάρμπα, έχουμε ακόμη έναν ε, συνάδελφο που θέλει το λόγο, κύριο Στάνοκ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Πριν από δύο χρόνια ζήτησα απαγόρευση πτήσεων, μια ζώνη απαγόρευση πτήσεων στο Κοινοβούλιο θα είχαν σωθεί δεκάδες χιλιάδες ζωές πιστεύω αν είχε γίνει αυτό εάν η Δύση είχε εφαρμόσει μια τέτοια στρατηγική. Αλλά τώρα το ερώτημά μου είναι το εξής. δεδομένου του καθεστώτος που παρία που έχει πετύχει η Ρωσία μετά τη συμπεριφορά της και την επίθεση κατά της Ουκρανίας, πιστεύετε ότι θα υπάρξει επίδραση στο πώς ε, τοποθετείται η Ουάσινγκτον ή οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και αμφισβητώντας πια τη στήριξη της Ρωσίας προς τον Ασάντ θα ξανασκεφτούν το θέμα της απαγόρευσης πτήσεων διότι η χρήση των ε, αυτοσχέδιων ε, βομβών ε, από παρέλια που οδηγούν στο θάνατο τόσων πολιτών είναι απαράδεκτο. Οι Αμερικανοί με τις προηγμένες τεχνολογίες που διαθέτουν και τους αντιπρευλακούς τα υπερβολικά του συστήματα θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν τα, τους πυράβλους του Αλασάτ και τις βόμβες του και να δημιουργήσουν μια ζώνη απαγόρευσης πτήσεων. Η Ρωσία είναι γνωστό ότι στηρίζει το βάρβαρο καθεστώς του Ασάντ, αλλά έχει ε, ε, εξεγείρει εναντίον της και τον υπόλοιπο πολιτισμένο κόσμο με τη συμπεριφορά της. Πιστεύετε λοιπόν ότι αυτό μπορεί να οδηγήσει σε πίεση και προς τον Ασάντ για να έρθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Τάνο. Ο κύριος Αλνταρμπά έχετε το λόγο. Απαντήστε παρακαλώ στις ερωτήσεις των ε, βουλευτών. Ε, Ευχαριστώ. Ευχαριστώ όλους και όλες που έθεσαν ερωτήσεις. Πρώτα απ' όλα για την ε, διεθνή απόκριση, την ευρωπαϊκή απόκριση προς την κρίση. Η απόκριση αυτή ήταν αρκετή, βεβαίως και όχι, ήταν ε, ανεπαρκής και βλέπετε το εύρος, τις διαστάσεις που έχει πάρει η ανθρωπιστική αυτή τραγωδία και το πόση βοήθεια χρειαζόμαστε το τι πολιτικά πλήγματα έχουμε δεχτεί και το ε, τι στατιωτική καταστροφή επίσης υπήρξε. Ξέρουμε ότι ήταν αξιέπαινη η στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μεν, αλλά εδώ μιλάμε για μια επανάσταση που στόχο έχει να κερδίσει την ελευθερία και για μια επανάσταση που έχει σκοπό να επιβεβαιώσει την πίστη μας προς αυτούς που μας στήριξαν. Επιβεβαιώνουμε λοιπόν και εμείς την πίστη και την ευγνωμοσύνη μας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση που προσπάθησε να μας βοηθήσει. Δυστυχώς όμως αυτή η βοήθεια δεν ήταν επαρκής. Ω προ τι διαπραγματεύσει τη Γενέβη, τέθηκαν κάποιε ερωτήσει. Θα απαντήσω συνολικά με μία και μόνη απάντηση. Γιατί η διαδικασία των διαπραγματεύσεων στη Γενέβη απέτυχε. Το γνωρίζουμε, είναι σαφές ότι απέτυχε. Γνωρίζοντας ότι ένα εγκληματικό καθεστώς κυβερνά τη Συρία και πώς συμπεριφέρεται, καταλαβαίνουμε ότι μία ειρηνική λύση δεν θα είχε γίνει αποδεκτή. Ε, το καθεστώς που σκοτώνει τους ε, πολίτες του με πυράβλους με πυράβλους Κουντ δεν είναι ένα ειρηνικό καθεστώς. Είναι ένα καθεστώς που επιτίθεται στους αμάχους που χρησιμοποιεί χημικά όπλα εναντίον τους. Και εμείς, η διεθνής κοινότητα, τι κάνουμε. Εγκρίναμε ένα ψήφισμα, ε, διεθνές μεν, αλλά για την απόσυρση, την ε, εξάλληψη των χημικών όπλων. Ε, ψηφίστηκε αυτό, εντάξει, αλλά επιτρέπουμε τα συμβατικά όπλα, τα κλασικά, τα γνωστά και παραδοσιακά όπλα να χρησιμοποιούνται κατά των σύρων πολιτών σε αντάλλαγμα. Τι θα πει, εξαλείπουμε τα χημικά για να επιτρέψουμε τα συμβατικά κατά του λαού της Συρίας που δολοφονείται καθημερινά. Να επανέλθω στο θέμα της Γενέβης. Ο στόχος των διαπραγματεύσεων στη Γενέβη ήταν να δημιουργηθεί μια μεταβατική κυβέρνηση ή έστω ένα συνασπισμός ε, για να οδηγήσει τη χώρα στην, ε, σε, κυβέρνηση, σε εκλογές. Ένα συλλογικό σώμα που θα μπορούσαν να υποβάλουν υποψηφιότητα πολίτες και στατιωτικοί και επί ένα-δυο χρόνια να ε, εξασφαλίσει την σωστή μετάβαση προς τις δημοκρατικές πια εκλογές ένας τέτοιος φορέας κυβερνητικός για να υπάρξει πραγματική μετάβαση σε επίπεδο εξουσίας ήταν απαραίτητο. Έπρεπε να υπάρχει όμως συμφωνία και από την αντιπολίτευση και από το επίσημο καθεστώς της Συρίας. Είπαμε τους Αμερικανούς, τους Ευρωπαίους, τους Ρώσους και τους ε, τους Άραβες ότι δεν μπορεί να δημιουργηθεί τέτοιο μεταβατικό καθεστώς διότι ε, το κυβερνών καθεστώς έχει ένα πράγμα στο μυαλό του ή Ασάντ ή φωτιά στα πάντα. Το κυβερνών λοιπόν καθεστώ δεν υπήρχε περίπτωση να δεχτεί τέτοιον ε, φορέα, ε, τέτοιο κυβερνητικό σχηματισμό έστω και προσωρινά, χωρίς τη συμμετοχή του Ασάντ. Επίσης υπάρχουν και ρωσικές πιέσεις, όπως είπατε, και στη Γενέβη μεταβήκαμε γνωρίζοντας όλες αυτές τις πληροφορίες. Είχαμε υπόψη ότι όλη η όλη διαδικασία δεν πρόκειται να καταλήξει σε κάποιο αίσιο αποτέλεσμα, σε πολιτική λύση αλλά ως προς την διαμεσολάβηση, ως προς τις διαπραγματεύσεις και τη διαπραγματευτική μας θέση, κερδίσαμε κάτι στη Γενέβη, διότι το ψήφισμα της Γενέβης 1, του πρώτου γύρου των διαπραγματεύσεων, έλεγε με σαφήνεια ότι δεχόμαστε την ειρηνική λύση. Δεχόμασταν τη λύση που πρότεινε η Γενέβη 1, δηλαδή την απόσυρση των στρατευμάτων, την επιστροφή τους στους στρατώνες τους και την ε, δυνατότητα να μπορέσει ο λαός να διαδηλώσει και να διαμαρτυρηθεί ειρηνικά. Διεκδικήσεις ε, που ε, ε, επικυρώνονταν από το ψήφισμα της Γενέβης 1. Εμείς το δεχτήκαμε το ψήφισμα αυτό. Και με την προσέλευσή μας στο δεύτερο γύρο των διαπραγματεύσεων, στη Γενέβη 2, δείξαμε ότι το καθεστώς Ε, ε, εξεφ, εκφράστηκε βάσει των λόγων του, των όσων είχε υποαγορεύσει ο κύριος Αλασάντ και τοποθέτησε ε, του Υπουργού Εξωτερικών της Συρίας απευθυνόταν μόνο στους ε, προσκύμενους τον κύριο Ασάντε. Εμείς απευθυνθήκαμε στον κόσμο ολόκληρο, σε όλους τους Σύρους. Είδαμε την αδιάλακτη στάση ενός επίσημου καθεστώτος. Εμείς πήγαμε στη Γενέβη ανοιχτόμυαλοι, καθίσαμε στο ίδιο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τους εκπροσώπους αυτού του καθεστώτος. Δεχτήκαμε να κάνουμε παραχωρήσεις, παρόλο που γνωρίζαμε ότι το κοινό μα και ο λαό τη Συρία δεν ήθελε να πάμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με το επίσημο καθεστώ και να διαπραγματευτούμε μαζί του. Όμω εμεί το κάναμε. Το πράξαμε και πήγαμε στη Γενέβη. Η κυρία ε, συνάδελφος βουλευτής που μίλησε για τη συνεργασία με τις φονταμενταλιστικές δυνάμεις και τους εξτρεμιστές ε, να σας πω ότι στη Γενέβη πήγαμε αφού συζητήσαμε με όλε αυτέ τι ομάδε, που σε κάποιε περιπτώσει είναι το δεξί μα χέρι στο εσωτερικό τη χώρα. Όλε αυτέ οι ομάδε μα ανέθεσαν την διαπραγματευτική εντολή να μιλήσουμε εξ ονόματό του. Πήγαμε λοιπόν στη Γενέβη και είχαμε πίσω μα την δική του στήριξη, καθώ και τη διάθεση να δεχτούμε εκεχηρία. Όμω αυτό που συνέβη στην Γενέβη είναι ότι το καθεστώς οδήγησε σε αποτυχία αρνήθηκε και ε, εξαφάνισε κάθε δυνατότητα εξέβρεσης πολιτικής λύσης. Αυτά για τη Γενέβη. Τώρα θα ήθελα να μιλήσω για την ε, ανάγκη να βρούμε ένα στάδιο που θα ακολουθήσει αυτό το κενό μετά τη Γενέβη. Μία διάσκεψη, μία διάσκεψη που όμως θα παραμένει κατά την άποψή μου εντός εισαγωγικών ορφανή. Ακριβώς λόγω της επίσημης θέσης του κυβερνώντος καθεστώτος. Δεν υπάρχει καμία διάθεση συνεργασίας από πλευράς τους. Ως προς την τρομοκρατία τέθηκε και ως προς αυτό ένα ερώτημα. Το τρίτο ερώτημα τέθηκε και άλλο ερώτημα, τέθηκαν πολλές ερωτήσεις καλύτερα για το θέμα αυτό, για τους εκτρεμιστές. Η δική μας θέση είναι σαφής. Σας ε, είχαμε πει ότι στις περιοχές που απελευθερώθηκαν από τις ελεύθερες φυλιακές δυνάμεις εδώ και ένα χρόνο ήρθαν ε, οι, εξτρεμ, οι εξτρεμιστικές αυτές ομάδες και μερικές φορές κατάφεραν να κερδίσουν και τον έλεγχο αυτών των περιοχών. Εμείς τους ε, αντιμαχόμαστε εδώ και ένα χρόνο. Είναι δυο λογιών αυτοί οι εξτρεμιστές. Είναι είτε φυλακισμένοι το επίσημο καθεστώτος που βγήκαν από τις φυλακές δραπέτευσαν ή είχαν αποσταλεί στο Ιράκ τη στιγμή της Αμερικανικής και Βρετανικής ε, παρέμβασης στο Ιράκ για να ρίξουν βόμβες, για δολιοφθορά και ούτω καθεξής. Οι φυλακισμένοι αυτοί λοιπόν απελευθερώθηκαν απελευθερώθηκαν για να ασκήσουν την βία τους στο εσωτερικό της χώρας. Η δεύτερη κατηγορία ήρθαν ε, έξωθεν είναι μέλη της Αλκάιντα πολλές φορές, προσκύμενοι στην Αλκάιντα και μερικές φορές έχουν έρθει και από ευρωπαϊκές χώρες. Θα πρέπει λοιπόν να έχετε όλοι υπόψη το εξής. Εμείς αγωνιστήκαμε κατά των εξτρεμιστών αυτών. Το καθεστώς το καθεστώς που μας ε, προσπάθησε να μας καταστήλει βία ε, και καταγγέλει τους εξτρεμιστές ουδέποτε τους πολέμησε. Εμείς τους πολεμήσαμε, τους πολεμούσαμε πάντοτε. Πριν το τέλος του 2013 οι στρατιώτες μας, οι αγωνιστές μας ξεκίνησαν μια πολύ βίαιη επίθεση, μια, μια προσπάθεια πολύ ε, σταθερή να αντιμετωπίσουν αυτούς τους ε, εξτρεμιστές από το Λίβανο λόγου χάρη σε μια σειρά από πόλεις της χώρας. Πρόκειται για εξτρεμιστές που τους ξέρουν όλοι. Υπάρχουν ε, αγωνιστές που έχασαν σαν μάρτυρες τη ζωή τους σε την την ε, δρυμία επίθεση κατά των εξτρεμιστών. Έχουμε δώσει λοιπόν ε, αγώνα ε, σε αγώνων για να αντιμετωπίσουμε τους εξτρεμιστές και παρόλα αυτά οι εξτρεμιστές παραμένουν οι καλύτεροι σύμμαχοι του κυβερνώντος καθεστώτος. Το ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι έχουμε κάνει πραγματική μάχη για να αντιμετωπίσουμε αυτούς τους τρομοκράτες όλοι, εμείς όλοι από την πλευρά του λαού της Συρίας και εσείς από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να, να πολεμήσουμε αυτούς τους δύο οργανισμούς και τους εκπροσώπους του Ισλαμικού κράτους της Μέσης Ανατολής, του Λεβάντε και τους υποστηρικτές του Αλασάντ που έχουν διαπράξει ένα σωρό βιαιότητες κατά του λαού της Συρίας. Τώρα, έγινε λόγος για μειονότητες, έγινε λόγος για τους χριστιανούς. Συγκεκριμένα, εγώ ανήκω σε μια, προέρχομαι από μια περιοχή, καταγωγή από μια περιοχή, όπου η πλειοψηφία είναι χριστιανή. Είναι η πόλη του Αλμισλή, όπου υπάρχουν ένα σωρό ε, χριστιανοί. Είναι μια πόλη που ιδρύθηκε από τους Γάλλους το 1921. Υπάρχουν χριστιανοί καθολικοί, προτεστάντες και ορθόδοξοι. Στην πόλη αυτή υπάρχουν Σύριοι με καταγωγή από τη Συρία, αλλά και αλλά και με πολύ παλιά ιστορική καταγωγή. Ε, είναι μια παλιά ε, μια παλιά Συριακή, πόλη της Συρίας αυτή. Τους ε, χριστιανούς τους δεχτήκαμε με ανοιχτές αγκάλες. Εγώ προσωπικά πήγα σχολείο σε ποτεσταντικό ε, σχολείο, από το δημοτικό έως ε, ε, το λύκειο. Μιλάμε για ένα σχολείο που δικούσαν προτεστάντες και στη δική μου την περίπτωση, στο δικό μου το σχολείο, αλλά και σε άλλα σχολεία της πόλης. Οι δάσκαλοι μου Οι τότε δασκαλοί μου είναι ακόμη στη Συρία και είμαι ακόμη σε επαφή μαζί τους. Ζήσαμε σε μια περιοχή, μια περιφέρεια, όπου δεν γινόταν κανένας διαχωρισμός μεταξύ Αράβων, Κούρδων, Χριστιανών, Μουσουλμάνων, σε μια περιοχή ήρεμη, ειρηνική, οι χριστιανή, Πριν τον ε, Μπασάρ, τον πατέρα του Μπασάρ, Είχαν εκκλησίες, μπορούσαν να χρησιμοποιούν ως σύμβολο το Σταυρό. Βεβαίως και μπορούσαν. Μετά την αποχώρηση των Γάλλων το 1946, μετά την αποχώρησή τους και ως το 1970, τι συνέβαινε, ποιο ήταν το καθεστώς των χριστιανών. Οι χριστιανοί, πολύ απλά, όπως και οι μουσουλμάνοι, μπορούσαν να ζήσουν όπως ήθελαν. Υπήρχε μια απόλυτη, μια διατάραχτη ειρήνη, ένα δημοκρατικό καθεστώς, με, κάποιες, βέβαια, με κάποιους αλλά πάντοτε η δημοκρατία περτερούσε. Οι χριστιανοί είχαν, τα ίσα, ίσα δικαιώματα με τους μουσουλμάνους, εκπροσωπούνταν στο κοινοβούλιο και εγώ γνωρίζω έναν πρόεδρο της Βουλής, ο κύριο, τον κύριο Σαϊτσάκ, ο οποίος ήταν χριστιανός ορθόδοξος και ήταν πρόεδρος της Βουλής στα... στις αρχές της του 50. Ήταν ένα από τα σύμβολα της Συρίας, ένας χριστιανός Σύρος χριστιανός που του οποίου η οικογένεια ήταν από αιώνες στη Συρία και ανήκε στην παράταξη που αντιμαχόταν την παρουσία της Γαλλίας στη Συρία. Ο μεγάλος μας οικονομολόγος, ο κ. Λαντακή, είναι ένας μεγάλος, ένας χριστιανός μάλλον, ο οποίος έχει παραμείνει μια από τις μεγαλύτερες μορφές της ιστορίας της Συρίας. Εγώ επτά μήνες μετά την Επανάσταση ε, έτυχε να πάω στην εκκλησία Μεγάλη Παρασκευή την περίοδο του Πάσχα και μίλησα με τον Πατριάρχη και των Ορθοδόξων και των Καθολικών και των ε, ε, προτεσταντών για να για να τους ευχηθώ για την ε, γιορτή αυτή, για το Πάσχα. Δεν υπήρχε λοιπόν καταπίεση των χριστιανών. Αυτά είναι ψεύδι. Ο πατέρας του Μπασαραλασάντ ε, ιδιοποιήθηκε αυτήν την εικόνα. Οι χριστιανοί ήταν γεωργοί, ζούσαν στην Ήπεθρο. Εκείνος όμως κατοικοποίησε όλες του, όλους τους βιομηχανικούς κλάδους, ακόμη και την αυτοκινητομηχανία και οι περισσότεροι χριστιανοί μετανάστευσαν. Μετανάστευσαν εκτός χώρας, στον Καναδά, στις Ηνωμένε Πολιτείες, σε χώρες του Βορρά και της Δύσης, από τον προηγούμενο αιώνα. Πρέπει λοιπόν όλοι να έχουν υπόψη ότι αυτό οι άνθρωποι αυτού του καθεστώτο είναι ψεύτε. Είναι ψεύτε γιατί δεν προστατεύουν τι μειονότητε. Ούτε τι μειονότητε. Οι μειονότητε και η πλειοψηφία προστατεύονται από τη δημοκρατία. Είμαστε σε μια χώρα που σέβεται κάθε μειονότητα, σέβεται την ανεξιθρησκεία. Ε, είχαμε ταχθεί ανέκαθεν κατά της τρομοκρατία και είμαστε υπέρ της ε, πολυφωνία αυτού του ψηφιδωτού που συνθέτει την σύγχρονη Συρία. Ούτε οι μειονότητε ούτε η πλειοψηφία τη Συρίας όμω μπορούν να συνεχίσουν να ζουν υπό τι σημερινέ συνθήκε. Βλέπω ότι η προπαγάνδα του επίσημου καθεστώτο έχει κερδίσει τελικά έδαφος και υποστηρικτές ιδίω ε, μεταξύ των δυτικών. Εγώ πραγματικά σας ε, θέτω σε επιφυλακή κατά της προπαγάνδας αυτής. Ζούμε μία μαύρη περίοδο στην ιστορία μας ε, τα τελευταία τρία χρόνια. Είναι ενωμένε όλες οι μειονότητες. Όταν εκτοξεύεται ένα πύραυλο, δεν γίνεται καμία διάκριση μεταξύ Αράβων ή Κούρδων, Χριστιανών ή Μουσουλμάνων. Είναι ένα πύραυλο που σκοτώνει τους πάντες, χωρίς να γίνεται διάκριση μεταξύ μειονοτήτων ή πλειοψηφία. Έχουμε και αποδείξεις. Εσείς αυτή τη στιγμή βρίσκεστε ενώπιον ενός μεγάλου ανθρωπιστικού εγκλήματος. 11.000 φυλακισμένοι θανατώθηκαν μέσα σε ένα σοφρονιστικό ίδρυμα. Έχετε εικόνες που τα αποδεικνύουν. Και το είπαμε 48 ώρες πριν ξεκινήσουμε και πραγματεύσεις στη Γενέβη 2. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα εγκλήματα τη τελευταία τριετία. Δείτε τι διαπράττει το καθεστώ αυτό ω έγκλημα. Σε ό,τι αφορά την Κίνα. Σε ό,τι αφορά την ε, Κίνα, συναντήσαμε εκπροσώπους της Κίνας στο Μοντρέ και μετά την ομιλία μας εκεί. Εγώ συνάντησα τον ε, Υπουργό Εξωτερικών Υποθέσεων της Κίνας, μια συνάντηση εξαιρετικά χρήσιμη, διότι εξέφρασε την κατανόησή του, αλλά είπε ότι η αντιπολίτευση σε κάποιο βαθμό σφάλει. Ταυτόχρονα όμως δήλωσε ότι τα όσα λέει ο πρόεδρος Μπασάρα Λασάντ είναι επίσης τελείως εσφαλμένα, είναι στην κακή κατεύθυνση, ενώ τουλάχιστον η αντιπολίτευση έχει θετική επικοδομητική προσέγγιση. Απίφθινε λοιπόν έκκληση και πρόσκληση για να επισκεφθούμε επισήμως την Κίνα και εγώ θα απαντήσω στην πρόσκληση αυτό προσεχώς. Έχουμε πολύ καλές σχέσεις με την Κίνα και τους ε, Κινέζους πολιτικούς Σε ό,τι αφορά τώρα το ερώτημα που τέθηκε για το Ιράν. Το Ιράν προσκλήθηκε επίσης δέχτηκε το ανακοινωθέν που προέκυψε από τον πρώτο γύρο διαπραγματεύσεων στη Γενέβη και επίσης δέχτηκε μία πρόσκληση την αποδέχτηκε συγκεκριμένα. Όμως δεν μπορεί κάποιος που δεν προσυπογράφει στο ανακοινωθέν της Γενέβης 1 να συμμετέχει στη Γενέβη 2. Το Ιράν συμμετείχε στις βιαιότητες της Συρίας, η Χεσμολάχ, που είναι μια τρομοκρατική οργάνωση δεν μπαίνει επισήμως στην Συρία, αλλά πιέζεται, πιέζεται από τους Ιρανούς. Η συμμετοχή λοιπόν στον πόλεμο της Συρίας μέσω της Χεσμολάρ δεν ε, είναι κάτι που το, βλέπει ευνοϊκά ο αραβικός κόσμος. Η Χεσμολάρ συμμετείχε λοιπόν σε αυτήν την ε, καταστροφή του Συριακού λαού και δεν δέχτηκε βεβαίως τη δήλωση της Γενέβης 1. Εάν το Ιράν θέλει πραγματικά να συμβάλλει επικοδομητικά στην εξέβρεση λύσης, εμείς το υποδεχόμαστε ε, χωρίς κανένα πρόβλημα. Ευχαρίστως να δεχτούμε την συμβολή τους. Όμως θα πρέπει προηγουμένως το Ιράν να φροντίσει οι εκπρόσωποι της εθνικής πολιτοφυλακής και της Χεσμολάχ στη Συρία να εξαλειφθεί. Θα πρέπει να δεχτούν την αναγγελία της Γενέβης 1. Γι' αυτό ακριβώς ακόμα αντιτιθέμεθα στη συμμετοχή του Ιράν στις διαπραγματεύσεις της Γενέβης. Σε ό,τι αφορά τώρα τις δυνάμεις της αντιπολίτευσης και το κατά πόσο ελέγχουμε τις δυνάμεις της αντιπολίτευσης. Βεβαίως, Πήγαμε στη Γενέβη έχοντας εντολή από όλες τις ε, ομάδες της αντιπολίτευσης. Και είμαστε αποφασισμένοι να στείλουμε βοήθεια σε όλες τις απελευθερωμένες ζώνες. Και οι ντόπιοι μαχητές ήταν το όπλο μας για την καταπολέμηση και την ανατροπή το καθεστώτος. Αυτοί οι αγωνιστές θα φροντίσουν να φτάσει η ανθρωπιστική βοήθεια σε όλους τους ήρους πολίτες. Μιλήσαμε για τη Γενέβη. το πείσμα του καθεστώτος Ασάντ είναι το μεγαλύτερο πρόσκομα, το βασικό πρόσκομα των διαπραγματεύσεων στη Γενέβη. Η αιμονή του. Με ρωτήσατε αν πιστεύουμε ότι μια στρατιωτική επέμβαση θα ήταν λύση. Όχι. Η λύση θα πρέπει να είναι πολιτική. Να βρεθεί πολιτική λύση. Βέβαια αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο παράλληλες γραμμές. Μία στρατιωτική και μία πολιτική και γνωρίζετε θαυμάσια ότι αν δεν ασκηθεί ισχυρότατη πίεση στο καθεστώς του Ασάτ δεν πρόκειται να βρεθεί πολιτική λύση. Όταν ε, χρησιμοποιήθηκαν χημικά όπλα μπροστά στα μάτια όλου του κόσμου ήρθα σε επαφή με τον Τζον Κέρι και άλλους υπουργούς εξωτερικών και όταν οι Ηνωμένε Πολιτείε, η Γαλλία και η Μεγάλη Βρετανία αντιτάχθηκαν στο καθεστώς και απείλησαν με στρατιωτική επέμβαση για να τιμωρήσουν τον Ασάντ για τη χρήση χημικών όπλων κατά του πληθυσμού, τότε μόνο υποχώρησε ο Ασάντ και συμφώνησε, συνθηκολόγησε να παραδώσει τα χημικά όπλα. Ιδού η απόδειξη ότι η μόνη γλώσσα που γνωρίζει αυτό το καθεστώς είναι η γλώσσα της βίας. Γιατί ανέκαθεν είχε στηριχθεί στη βία και μόνο τη βία καταλαβαίνει. Οπότε έχουμε, επαναλαμβάνω, δύο παράλληλες γραμμές. Μία πολιτική και μία στρατιωτική. Η στρατιωτική ισορροπία φυσικά επί τόπου στη Συρία θα πρέπει να κλείνει, και να κλείνει υπέρ των δυνάμεων της αντιπολίτευσης. Μόνο έτσι θα βρεθεί πολιτική λύση. Εμείς πρεσβεύουμε μια πολιτική λύση. Βέβαια, ένα τρίτο της χώρας έχει καταστραφεί, αλλά θεωρούμε ότι θα πρέπει να βρεθεί πολιτική λύση. Γι' αυτό όμω χρειαζόμαστε στρατιωτική δύναμη για να εξουδετερώσουμε τις, τη στρατιωτική αεροπορία του καθεστώτος. Και αν ασκηθεί πίεση στην πρωτεύουσα, στη Δαμασκό, τότε θα εξαναγκαστεί το καθεστώς να συμφωνεί σε μια πολιτική λύση. Θα ήθελα πάντως να σας καθησυχάσω και να σας διαβεβαιώσω ότι δεν θα πρέπει να φοβάστε ότι αν δώσετε όπλα θα πέσουν στα χέρια των τρομοκρατών και των εξτρεμιστών στη Συρία. Γιατί είμαστε ικανοί να καταπολεμήσουμε τους τρομοκράτες και τους εξτρεμιστές. Δεν θα βρεθούν στο πολιτικό προσκήνιο, θα αποκλειστούν από την πολιτική σκηνή. Γιατί οι πραγματικοί επαναστάτες ε, και αυτοί που θα καταπολεμήσουν τον Μπασάρα Σάντ είναι όλοι όσοι δίνουν, όσοι γίνουν το αίμα του σήμερα για τη Συρία. Εμείς ε, καταπολεμήσαμε τους Ισλαμιστές ε, και είμαστε κατά των Ισλαμιστικών δυνάμεων και του Ιράκ και άλλων χωρών. Δεν θα επιτρέψουμε σε κανένα να καπηλεθεί και να σφετεριστεί την επανάστασή μας. Είμαστε υπεύθυνοι για τις δηλώσεις μας. Όλοι όσοι είναι υπέρ των εκλογών, πραγματικών δημοκρατικών εκλογών ε, με προσέλευση της κάλπης ε, μας βρίσκουν Σε Αυτή τη γραμμή στηρίζουμε. Είμαστε υπέρ δημοκρατικών εκλογών. Υπάρχουν εθνοτικές διαφορές, υπάρχουν κοινοτικές διαφορές. Εφόσον όμως όλοι οι εκπρόσωποι των ομάδων είναι υπέρ δημοκρατικών εκλογών και σεβαστούμε τα αποτελέσματα των εκλογών, εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να συμμετέχουν όλοι σε μια δημοκρατική διαδικασία. μια γνήσια και δίκαιη πολιτική λύση θα πρέπει να επικρατήσει. Συμφωνούμε με τις συζητήσεις στη Γενέβη και όταν δεχτήκαμε την ε, σύσταση ενός ε, μεταβατικού φορέα, μιας μεταβατικής κυβέρνησης που θα παρτίζεται από μετριοπαθείς και από προσωπικότητες που θα ε, είναι αποδεκτές και από το καθεστώς και από την αντιπολίτευση. Ουσιαστικά δώσαμε το πράσινο φως για μια τέτοια μεταβατική περίοδο ώστε να περάσουμε σε μια πραγματική νέα δημοκρατική Συρία μετά τη διεξαγωγή δημοκρατικών εκλογών. Στη Συρία, όπως είπα και προηγουμένως, είμαστε μάρτυρες μιας ανθρωπιστικής τραγωδίας. Μια απαγόρευση πτήσεων λοιπόν μια ζώνη απαγόρευσης πτήσεων είναι αδιανόητη. Δεν είναι βιώσιμη μια τέτοια λύση. Δεν μας βρίσκει σύμφωνος. Είχαμε ζητήσει την απαγόρευση πτήσεων, αλλά στην πρώτη φάση της σύγκρουσης. Αλλά η συνένοχη σιωπή της παγκόσμιας κοινότητας συνέβαλε σε μια επιδείνωση της κατάστασης. Και σήμερα χρειαζόμαστε όπλα για να αντιμετωπίσουμε την πολεμική αεροπορία του καθεστώτος. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ανθρωπιστική βοήθεια, είδατε τον τεράστιο αριθμό των δολοφονιών. Έγιναν μαζικές δολοφονίες και εντός των φυλακών, αλλά και εκτός των φυλακών. Δολοφονίες αμάχων, γυναικών και παιδιών. Οι γυναίκες διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στη Συριακή Επανάσταση. Έπαιξαν πραγματικά ένα ηρωικό ρόλο. Βέβαια, ίσως να μην αναδείξαμε δεόντως ή να μην αναγνωρίσαμε όπω έπρεπε το ρόλο των γυναικών στην Επανάσταση. Πήγα στην πόλη Χαρά, στην ε, Συρία, την πόλη από την οποία ξεκίνησε η Επανάσταση και παρακολούθησα τις προσευχές στις μουσουλμανικές γιορτές. Συνάντησα μία γυναίκα ε, που καθόταν δίπλα στο παιδάκι της που είχε κατάγματα στα πόδια. Η γυναίκα αυτή μου είπε «Έχω δύο-τρία παιδιά που έχασαν τη, ζωή τους ως μάρτυρες και το τέταρτο παιδί μου είναι τραυματισμένο. Αλλά αυτό είναι το τίμημα που καλούμαστε να πληρώσουμε για την ελευθερία και τη δημοκρατία. Είναι πραγματική αυτή η ιστορία που σας διηγούμε. Αυτή η γυναίκα δέχτηκε να θυσιάσει τα παιδιά της για την ελευθερία της πατρίδας της. Για την ελευθερία της Συρίας. Αυτός είναι ο ρόλος που έπαιξε η, η μάνα στη Συρία, η γυναίκα μάνα στη Συρία. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη δημοκρατία. Έγινα πρόεδρος του Εθνικού Συνασπισμού των Συριακών Επαναστατικών και Αντιπολιτευτικών Δυνάμεων μετά από εκλογές. Θέλησαμε να δώσουμε το καλό παράδειγμα. Έχουμε πρόεδρο, αντιπρόεδρο, γενική γραμματέα, πολιτική επιτροπή. Όλα αυτά τα όργανα και οι επικεφαλείς τους ε, εξελέγησαν με δημοκρατικές ε, εκλογές. Αυτό είναι ο τρόπος που θα ακολουθήσουμε και για την σύνταξη του συντάγματος της Συρίας στο μέλλον. Θεωρώ ότι απάντησα στις απορίες σας, κάλυψα τις ερωτήσεις που μου θέσατε. Μου δώσατε πραγματικά μια μοναδική ευκαιρία να συναντήσω εδώ τα μέλη της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, γιατί θεωρούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο καλύτερος μας σύμμαχος, ο πλησιέστερος μας σύμμαχος και θα ήθελα να συζητήσουμε να σταθείτε στο πλευρό μας και όχι στο πλευρό των δολοφόνων. Η Ευρώπη ήταν ανέκαθεν με το πλευρό των θυμάτων. Η Ευρώπη ουδέποτε δεν υποστηρίξε τους θύτες, τους δημίους και ποτέ δεν θα το κάνει. Αυτή είναι και η ελπίδα μας. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσίαση αυτή, για τις εξηγήσεις σας. Σας υποστηρίζουμε ένθερμα, αλλά γνωρίζουμε ποιες είναι οι δυνατότητές μας και αν θέλετε και η κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε που δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα δεδομένης της φρικτής κατάστασης των θυμάτων, των προσφύγων, των εσωτερικά εκτοπισμένων. Ήμουν στο Λίβανο πρόσφατα. Ένα εκατομμύριο πρόσφυγες από τη Συρία. Ε, οικογένειες με παιδιά, γυναίκες χωρίς τους άντρες τους με τα παιδιά. Είναι πραγματικά ε, μια τεράστια καταστροφή. Και γι' αυτό λοιπόν ελπίζουμε όλοι πολύ σύντομα να φτάσουμε σε μια ειρηνική λύση προκειμένου ο κόσμος στη χώρα σας να μπορέσει να ζήσει ειρηνικά και με σωστή συνύπαρξη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Okay, so, Soll Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να σας καλέσω να στραφούμε στο επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη και θα έχουμε ανταλλαγή απόψε με τον James Moran, επικεφαλής της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Αίγυπτο. Η κατάσταση στην Αίγυπτο ε, είναι πλέον σε ένα κρίσιμο σημείο σε ό,τι αφορά το Σύνταγμα. πολλά θετικά σημεία συμπεριλαμβάνονται. Το θέμα είναι τι θα γίνει με τα ζητήματα εφαρμογής και για τα πολιτικά ζητήματα και για τα θέματα θεμελιωδών δικαιωμάτων, κατά πόσον θα εφαρμοστεί όντως ε, η ουσία του συντάγματος ή κατά πόσον πρόκειται για μία ε, πρόσωψη και μόνο. Ξέρουμε ότι ο πρόεδρος Μόση δεν κατάφερε να ανταπεξέλθει στις προσδοκίες της δημοκρατικής και ότι προσπαθεί να εκπροσωπήσει ένα τμήμα μόνο του Αιγυπτιακού λαού. Ελπίζουμε η μεταβατική κυβέρνηση να μην διαπράξει περαιτέλω σφάλματα Μουμπάρακ δύο πλήν, αλλά πραγματικά να ακολουθήσει το δρόμο του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας σε μια χώρα που υπάρχει και μειονότητα χριστιανική και ε, λοιπόν έτσι διαμορφώνεται η κατάσταση, έχει επιδεινωθεί περαιτέρω η κατάσταση δε επειδή η κατάσταση της Αττικής Αραβίας και των κρατών του Περσικού κόλπου και της αδελφότητας των μουσουλμάνων ε, έχει ανακηρυχθεί ε, τρομοκρατική οργάνωση αυτό λοιπόν ερωτιόμαστε τι επιρροή θα έχει τις επόμενου μήνες και τις επόμενες εβδομάδες δεδομένη και τη ιδιαίτερη κατάσταση και τη βίαιη κατάσταση που επικρατεί στην Αίγυπτο. Ελπίζουμε λοιπόν να υπάρξει αυτή η δυνατότητα για μια προελιστική κοινωνία και θα θέλαμε να ακούσουμε πώς εκτιμάτε και εσεί την κατάσταση. Κύριε Πρεσβευτά, έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, και καλή σας μέρα αξιότιμοι κυρίες και κύριοι. Θα βάλω τα δυνατά μου για να σας κάνω μία επισκόπηση κατάστασης της κατάστασης στο Καΐρο. Ε, σπάνια είναι έθριος ο ουρανός στο Κάιρο, ξέρουν όσοι το επισκέφτονται και δεν ε, υπάρχει διαφορά τώρα. Όπως ξέρετε, ετοιμάζεται το, το Σύνταγμα. Βέβαια, η εκστρατεία υπέστη το, το πλήγμα, το μποϊκοτάρισμα από την Συμμαχία για τη Δημοκρατία και δεν ήταν και πολύ ενθαρρυντικό και πρόσφερο το έδαφος ε, για τη, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Πάντως, ε, το ίδιο το έγγραφο, όπως είπε ο Πρόεδρος, ε, το σχέδιο του Συντάγματος περιλαμβάνει κάποια θετικά στοιχεία. Για παράδειγμα, ε, μερικές από τις ε, διατάξεις, ε, τις πιο προοδευτικές που περιέλαβε το Σύνταγμα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες και μια ισότητα των δύο φύλων είναι πολύ καλά. Βέβαια θα πρέπει αυτά για να γίνουν αποτελεσματικά να μετατραπούν σε εσωτερική νομοθεσία. Και θα δούμε και τα αποτελέσματα μετά τις προεδρικές εκλογές και τις βουλευτικές και θα δούμε Ποιε είναι οι νομοθετικέ διατάξει επίση υπάρχουν κάποιε διατάξει για, για τη διάκριση των εξουσιών, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την προεδρική εξουσία και την νομοθετική εξουσία. Προ, προτείνεται καλύτερη και ισχυρότερη νομοθετική εξουσία για την αντιστάθμιση της εκτελεστικής και μετά τη σύσταση της Βουλής, τη συγκρότηση της Βουλής, θα εξασφαλιστεί, πιστεύω, μια πιο ισορροπημένη διακυβέρνηση μεταξύ νομοθετικής και εκτελεστική εξουσία. και ελπίζω να ανανεωθεί και να αναζωογονηθεί η συνεργασία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Αιγυπτιακής Βουλής μετά τη συγκρότησή της. Και πολλοί πρώην και νυν βουλευτές της Αιγύπτου μου λένε πώς προσβλέπουν σε τέτοια συνεργασία και αναζωογόνηση συνεργασίες με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το συντομότερο δυνατόν. Το Σύνταγμα περιλαμβάνει και κάποια πιο επίμαχα σημεία όπως την υποβολή προσαγωγή πολιτών σε στρατιωτικά δικαστήρια. Αυτό είναι προβληματικό. Υπάρχουν όμως κάποια στοιχεία που ίσως χαράξουν το δρόμο για την επαναφορά της Αιγύπτου στη δημοκρατία. Τώρα, ε, ο εκλογικός νόμος μόλις έχει εκδοθεί υπήρχε ένα πρόβλημα γιατί δεν προβλεπόταν διαδικασία προσφυγών. Προς το παρόν δεν έχει διορθωθεί αυτό το πρόβλημα και δεδομένου το χρονοδιαγράμματος ε, που προβλέπει ε, το Σύνταγμα για τις προεδρικές εκλογές ε, μάλλον θα γίνουν το νωρίτερο το Μάιο. Ο Χάμπτιν Σαμπάχη που θα θυμάστε ήταν στον πρώτο γύρο με 21% των, των εκλογών του 2011. Δήλωσε ότι θα είναι υποψήφιο και στις επόμενες ε, προεδρικές εκλογές. Μάλλον ε, θα ε, συμμετέχει και ο κύριος Ασίσιος υποψήφιος, ε, υπουργός άμυνας, αλλά τα προγράμματά τους στα προεκλογικά δεν τα γνωρίζουμε. Θα περιμένουμε την έναρξη της προεκλογικής εκστρατείας. Βέβαια, όσο πλησιάζουμε προς εκλογές ε, δραστηριοποιούνται διάφορα κόμματα, ακόμη και τα Ισλαμιστικά. Το κόμμα των αδελφών μουσουλμάνων, το κόμμα της ε, Ελευθερίας και Δικαιοσύνης ε, δεν έχει υιοθετήσει σαφή ακόμη θέση. Πάντως το βέβαιο είναι ότι αυτή τη στιγμή η χώρα δεν φαίνεται να είναι έτοιμη για επανασυμφιλίωση. Ακόμη και αν μερικοί έγκυροι πολιτικοί και Αλμούσα πρόσφατα δήλωσαν ότι ίσως κάποια στιγμή θα ήταν σκόπιμο να επανέλθουν στη διαδικασία επανασυμφιλίωσης. Όλα αυτά λοιπόν ε, λαμβάνουν χώρες σε ένα περίπλοκο ε, προσκήνιο ε, απειλών, στην ασφάλεια και στη Χερσόνησο Σίνα και στην ενδοχώρα με πολλές διαδηλώσεις αλλά και με κινητοποίησεις και κοσμικών οργανώσεων και φυσικά με μεγάλη παρουσία των δυνάμεων ασφαλείας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδίκασε απερίφραστα και μάλιστα και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το ίδιο, όλες τις ε, τρομοκρατικές ενέργειες και τη χρήση βίας και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Έχουμε σοβαρές ανησυχίες ε, και για τα αποτελέσματά του στην Αίγυπτο, αλλά και για στην ασφάλεια γενικώ, ακόμη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί είχαμε σημαντικέ ε, αναταραχέ και μάλιστα η επίθεση σε ένα τουριστικό λεωφορείο στον Ταμπάπ τον περασμένο μήνα που πολλοί άνθρωποι έχασαν τη ζωή του ε, και ο οδηγό του ίδιου, ίσω ξεκινήσει μια νέα φάση στην ε, προεκλογική εκστρατεία. Γιατί θα επηρεάσει και τον τουριστικό κλάδο που ούτω ή άλλω έχει υποστεί πλήγμα. Γιατί εκατομμύρια άνθρωποι που εξαρτώνται από τον τουρισμό έχουν υποστεί το πλήγμα της δραστικής μείωσης ε, του τουρισμού τον τελευταίο καιρό. Επίσης, ε, η πολιτική διαδικασία θα πρέπει να είναι ανοιχτή σε όλους όσους καταδικάζουν τη βία και στερνίζονται τις δημοκρατικές αρχές και θα πρέπει αυτή η διαδικασία να είναι όσο πιο περιεκτική γίνεται, να μην αποκλεί κανέναν, όχι μόνο χάρη δημοκρατικής μετάβασης, αλλά και για μία μακροπρόθεσμη και βιώσιμη ασφάλεια. Γιατί σε αυτό προσβλέπουν οι Αιγύπτιοι πάνω απ' όλα μετά από όσα πέρασαν τα δεινά από τον Ιανουάριο του 2011. Προσβλέπουν στην ασφάλεια. Αυτό προσδοκούν. Και φυσικά θα πρέπει να ληφθούν υπόψη ανησυχίε για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Γιατί σίγουρα η ασφάλεια είναι το πρώτο ζητούμενο, αλλά σίγουρα κάποιε δράσει που έγιναν για την προστασία τη ασφάλεια ήταν υπερβολικέ. Και μάλιστα είχαμε το πρόσφατο ψήφισμα του ε, Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τα συμπεράσματα του Υπουργείου Εξωτερικών του περασμένου μήνα με αυτές τις ανησυχίες. Ε, μας ε, ενδιαφέρουν και οι διαδικασίες ε, διαλεύκασης παλιών εγκλημάτων. Ελπίζουμε να επισφευστούν οι διαδικασίες. Πάντως μας ανησυχούν αυτές οι διαδικασίες. Επίσης, δίκες δημοσιογράφων, κάποιες καταδίκες διαδηλωτών που κατά τη γνώμη μας ήταν υπερβολικές, δυσανάλογες και φυσικά οι συνθήκες που μας ανησυχούν όχι μόνο για τους Ισλαμιστές αλλά και για εκπροσώπους κοσμικών οργανώσεων που επίσης φυλακήθηκαν. Ο Σταύρος Λαμπρινίδης σας ενημερώνει για τα θέματα αυτά. Ήταν πριν από λίγες εβδομάδες στο Κάιρο και συναντήθηκε με εκπροσώπους τη κυβέρνηση και της κοινωνίας των πολιτών και μαζί με τις αποστολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Κάιρο παρακολουθούμε εκ του κατά την κατάσταση και στη δική μας αντιπροσωπεία. Κύριε Πρόεδρε, αναφερθήκατε στους χριστιανούς. Νομίζω ότι η κατάσταση των χριστιανών βελτιώθηκε κάπω τους τελευταίου μήνε, μετά από ένα πολύ δύσκολο 2013 με εμπρισμούς εκκλησιών, οπότε έχουμε αρκετέ ισοδοξίε για τη θέση των χριστιανών στη χώρα. Περνάμε τώρα στην οικονομική πολιτική. Εκεί υπάρχουν κάποια ενδεικτικά σημάδια και μάλιστα ο Ιμπραήμ Μαχλέπ και η κυβέρνηση ε, ε, διόρισε σημαντικούς ε, οικονομολόγους στην κυβέρνηση που είναι πολύ πιο εμπειρογνώμονες σε θέματα οικονομικά. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί η Αίγυπτος εξαρτάται από τη γενεοδορία τριών χωρών του Περσικού κόλπου. Αυτό βέβαια δεν θα συνεχίσει στο μέλλον και το δήλωσαν ήδη δύο από τις χώρες του κόλπου. Οπότε χρειάζεται ευρύτερη υποστήριξη η Αίγυπτος ε, και με τεχνογνωσία και παροχή συμβουλών, αλλά πρέπει πρώτα να διεκπαιρεωθεί η διαδικασία των εκλογών. Και μάλιστα ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Αλσίση και ο Υπουργός Οικονομικών ε, τόνισαν ε, ε, πόσο έθρευστη είναι η πολιτική και πόσο τροτές είναι οι πολιτικές και έδωσαν έμφαση στο πρόβλημα των ε, επιδοτήσεων καυσίμων που είναι το 20% του προϋπολογισμού, 10% του ΕΕΠ και δημιουργεί τεράστιες ε, προκλήσεις για την οικονομική ανάπτυξη. Χρειάζεται μεγαλύτερο συντονισμός και μια διαδικασία αφύπνης και συνειδητοποίησης και φυσικά μια μεταρρύθμιση των επιδοτήσεων. Ε, προτείνεται αύξηση των φόρων, ε, πολύ πιο ρεαλιστικές προβλέψεις, ε, παρόλο που θα υπάρχει αύξηση του προπολογισμού κατά 12% φέτος, προτείνονται μεταρρυθμίσεις και στην ενεργειακή πολιτική, μεγαλύτερο άνοιγμα. Φαίνεται ότι γίνονται βήματα προς σωστή κατάθεση και προς μεταρρυθμίσεις. Και ε, υπουργοί με οικονομικά χαρτοφυλάκια για επενδύσεις, εμπόρια κτλ έχουν δείξει πολιτική βούληση να βελτιώσουν το επιχειρησιακό το επιχειρηματικό πνεύμα στην Αίγυπτο που έχει πληγεί τα μάλα τα τελευταία δύο χρόνια και επιτέλους ε, υιοθετήθηκε το νομοσχέδιο για τις επενδύσεις και μετά που θα εφαρμοστεί θα εξασφαλιστεί η ασφάλεια δικαίου για τις συμβάσεις και για τις επενδύσεις γιατί πολλές ευρωπαϊκές επιχειρήσεις επλήγησαν από την αβεβαιότητα αυτή κυρίως ε, μετά από ιδιωτικοποίησεις ε, ήταν πραγματικά σοκ ε, και φοβερή αυτή η κραδασμή για τους επενδυτές και χαίρομαι που η κυβέρνηση θα το αντιμετωπίσει αυτό. Βέβαια βρισκόμαστε ακόμη πρόωρη φάση και δεν ξέρουμε πόσο θα, κατά πόσο θα μακροημερεύσει αυτή η κυβέρνηση. Έχουμε τον τέταρτο πρωθυπουργό που τα έλαβα εγώ τα καθήκοντά μου, οπότε Ελπίζω να καταφέρει η κυβέρνηση να διεκπαιρώσει αυτά που ξεκίνησε, αλλά θα το δούμε, δεν είναι σίγουρο. Πάντω ήδη έχει ξεκινήσει μια κατεύθυνση προ μεταρρυθμίσει ε, και έχουν δρομολογηθεί. Πολύ καλό και ενθαρρυντικό. Τώρα για εξωτερική πολιτική έχουμε αρκετέ εξελίξει, αλλά δεν έχουμε χρόνο να τι αναλυσουμε ολε όλες. Μία-δύο θα σα αναφέρω επιγραμματικά. Η νέα σχέση, η αναζωογονημένη σχέση τη Αιγύπτου με την Ρωσία έχει σημειωθεί. Έγιναν σημαντικές επισκέψεις υψηλού επίπεδου για την αναζωγόνηση αυτής της σχέσης. Ίσως συνδέεται με την ε, αναδιάταξη, ανακατάταξη της ε, αιγυπτιακής εξωτερικής σχέσης ε, στον κόσμο. Η Ρωσία ενδιαφέρεται και η το συγγνώμη ενδιαφέρεται για την αναζωγόνηση των σχέσεών της με τις αφρικανικές χώρες. Καλό είναι να δημιουργηθεί μια να δημιουργηθούν γέφυρες ε, με την Αφρικανική Ένωση. Υπάρχει πρόβλημα όμως με τα νερά του Νείλου και το φράγμα της ε, κατασκευή φράγματος στην Αιθιοπία. Βέβαια είναι κάπως θεταμένη σχέση με την Αιθιοπία αυτή τη στιγμή. Ίσως εκεί χρειαστεί κάποια βοήθεια από παγκόσμιους φορείς όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάντως Είπαμε ότι αν ζητηθεί στήριξη θα πρέπει να ζητηθεί και από τις δύο πλευρές και η Αιθιοπία δεν φαίνεται να ενδιαφέρεται αυτή τη στιγμή. Φαίνεται ότι αυτό το θέμα θα μπορούσε να προκαλέσει πολιτικές δυσκολίες στις επόμενες μήνες τέλος και να στραφώ στις δικές μας δεσμεύσει. Κύριε Πρόεδρε, όπως τα γνωρίζετε, η Ευρωπαϊκή Ένωση για πρώτη φορά ε, από την Ευρωπαϊκή Ένωση ζητήθηκε να κινητοποιήσει για πρώτη φορά ε, αποστολή παρακολούθησης των εκλογών για τις ε, προεδρικέ ε, εκλογέ και έχουν ξεκινήσει προετοιμασίε και ασφαλώ. θα είναι πάρα πολύ σημαντικό να ε, ελεγχθεί εντελεχώ η διεθνής νομοθεσία για τις εκλογές και να παρακολουθηθεί ιδιαίτερω η εκστρατεία, η προεκλογική, δεδομένου και του δύσκολου περιβάλλοντος που επικρατεί ήταν δύσκολο ε, όταν ακούσαμε πριν από κάποιες εβδομάδες όταν ο κ. Λαπρινίδης ήταν εκεί από υψηλούς αξιωματούχους και στον τομέα της ασφάλειας ότι θα γίνει ό,τι είναι δυνατόν για να είναι ίσες οι συνθήκες ε, για τους ε, υποψηφίους. Άρα όσο πιο γρήγορα επιβεβαιωθεί η ημερομηνία για τη διεξαγωγή των εκλογών, γιατί δεν υπάρχει ακόμα η ημερομηνία αυτή, τόσο πιο γρήγορα θα ξεκινήσουμε την ανάπτυξη των δυνάμεων μας, της αποστολής μας. Είναι λοιπόν θετικό το γεγονός αυτό και θεωρώ ότι θα εμβαθύνει τις σχέσεις μας και θεωρώ και τον αμοιβαίο σεβασμό μας. Νομίζω ότι το επίπεδο πολιτικής δέσμευσης της ε, Λέδης Άστον εξακολουθεί να παραμένει υψηλό. Έξι φορές επισκέφθηκε την ε, χώρα. Ο Μπενεδίνο Λιά είναι τόσο συχνός ε, επισκέπτης. Έρχεται να φέρει και στο Κοινοβούλιο τα αποτελέσματα των εργασιών του που θεωρώ ότι θα πρέπει να το φιλοξενώ κάθε φορά που έρχεται. Και φυσικά θα πρέπει να βελτιώσουμε τις προσπάθειές μας για να υποστηρίξουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα και την κοινωνία των πολιτών, είτε με οικονομική βοήθεια, είτε με κίνητρα. Είναι πολύ ευαίσθητο το θέμα της ε, ξένης επιρροής ε, σε εισαγωγικά. Αν θέλουμε λοιπόν να υπάρχει ε, αποτελεσματικότητα θα πρέπει και από τις δύο πλευρές να υπάρξει καλή συνεργασία, καλέ νομοθετικέ πρακτικέ, για παράδειγμα. Εδώ πέρα σε αυτό το σημείο μπορεί να συμβάλλει τα μάλλα το δικό, μα το δικό σα το κοινοβούλιο. Ελπίζω λοιπόν να υπάρξει μεγαλύτερη δέσμευση για το μέλιο. Ο κ. Λαμπλινίδης θα συνειδητοποιεί αυτό απόλυτα και ενώ κάνει τη δουλειά του σε ό,τι αφορά την ε, εκπροσώπηση, εξακολουθεί να προσπαθεί να βελτιωθεί το νομοθετικό πλαίσιο σε ό,τι αφορά την αρρωγή και την πολιτική γειτονία. Οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Εξωτερικών τόνισαν ότι θα συνεχίσουν να υποστηρίζουν την οικονομική ανάπτυξη στην, ε, της κοινωνίας των, πολιτών. Και είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι την προηγούμενη εβδομάδα παρουσιάστηκε νέος χάρτης για την ένδυα στην Αίγυπτο και το ποσοστό έχει αυξηθεί από το 21% το 2010 σε 26% σήμερα το ποσοστό ένδυο προκαλεί ασφαλώς ιδιαίτερες ανησυχίες και ασφαλώς είναι οι νέοι, οι ευάλωτες ομάδες, οι γυναίκες, οι αγρότες που πλήττονται πιο πολύ. Άρα τα προγράμματα εστιάζονται σε θέματα απασχόλησης ε, για τους νέους, ε, εκπαίδευση, αστική ανάπτυξη και υπάρχουν σχέδια να γίνουν και πιο πολλά σε ό,τι αφορά τους λιγότερο ευνοημένους. Επίσης, ε, εξακολουθούμε να υποστηρίζουμε τις ε, χρηματοδοτήσεις από την Διεθνή Τράπεζα, από την Τράπεζα Επενδύσεων, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, μέσω της Ευρωπαϊκής Διευκόλυνσης και νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει σχετικές προτάσεις για χρηματοδότηση μέσα στην εβδομάδα. Σε ό,τι αφορά το εμπόριο και τι επενδύσει, έχουμε την ε, ε, βαθιά συμφωνία ελεύθερου εμπορίου, αν και ε, σε αυτή τη φάση αυτό που μετράει είναι η πολιτική συνέχεια και ίσως θα δούμε λοιπόν πώς θα διαμορφωθεί η κατάσταση μετά τις εκλογές. Καταλαβαίνουμε λοιπόν τις ε, δυνατότητες και τα πρώτα, τις πρώτες ενδείξεις που δείχνει η κυβέρνηση για την παροχή κινήτρων για το επιχειρηματικό Είναι θεραντικά αυτά. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητά μέλη, είναι σαφές ότι η Αίγυπτος είναι μια χώρα μεγάλης σημασίας για μένα. Σε Τρία χρόνια μετά την Επανάσταση υπάρχουν πάρα πολλές προκλήσεις ακόμα. Ο κατάλογος είναι πραγματικά πάρα πολύ μακρύ σε ό,τι αφορά τις λύσεις που μπορούν να εξευρεθούν μόνο στην Αίγυπτο την ίδια. Και ενώ μπορεί συχνά να μην συμφωνούμε, είναι από τους πιο παλιούς και τους πιο σημαντικούς εταίρους μας η εμπειρία μας σίγουρα μπορεί να τους βοηθήσει. Ε, το Κοινοβούλιο, και εδώ θα κλείσω κύριε Πρόεδρε, είναι ε, μεγάλος παράγοντας και πραγματικά αναμένω και ελπίζω να δω πολλούς από εσάς στο κάρο τους επόμενους μήνες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ όλοι ο Πρόεδρος. Κύριε Σαλαφρανκά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καλώς ήρθατε κύριε Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας σήμερα το πρωί και ευχαριστούμε για την πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση της κατάστασης στην Αίγυπτο. Την τελευταία φορά που επισκέφτηκα την Αίγυπτο ήταν ε, με την αφορμή μιας ε, task που διοργανώθηκε από την το πρόσωπο και έκτοτε βέβαια τα πράγματα έχουν αλλάξει πολύ. Ανησυχούμε με αυτή την κατάσταση αστάθεια στην Αίγυπτο, το είπατε κι εσείς, Υπάρχουν σοβαρές οικονομικές ε, αναταράξεις παρόλο που το έλλειμμα έχει περιοριστεί στο 12%. Η κατάσταση όμως είναι ανησυχητική. Το ποσοστό φτώχειας διαρκώς αυξάνεται στη χώρα αυτή. Το νομοσχέδιο που έχει στόχο να τονώσει τις, τις επενδύσεις είναι κάτι που παρόλα αυτά προτείνεται μέσα σε ένα κλίμα αναταραχών. Η επίσκεψη του κυρίου Ιλμπής, υπεύθυνο του παρατηρητηρίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ήταν ε, πολύ διαφανταστική για την κατάσταση στη χώρα. Όμως από τη δική σας την σκοπιά μας είπατε ποια είναι η άποψή σας για τις εξελίξεις στην ε, Αίγυπτο. Ξέρετε ότι για τη συνταγματική μεταρρύθμιση ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση απέστειλε μια αντιπροσωπεία για να παρακολουθηθεί μια όλη αυτή διαδικασία, όχι βεβαίως για τις επικείμενες εκλογές προεδρικές και βουλευτικές. Απλώς ήθελα να μου πείτε αν είστε σε θέση να μας δώσετε κάποια στοιχεία που να σχετίζονται με αυτή την έκθεση. Έκθεση που θα, μπορούσε, έκθεση που θα προκύψει ούτως ή άλλως από αυτή την υποστηρικτική αποστολή. Επίσης είπαμε ότι θα διεξαχθούν προεδρικές και βουλευτικές εκλογές. Εκλογές σε κλίμα πολυφωνίας και δημοκρατικής συμμετοχής. Οι δημοκρατικές και πολιτικές δυνάμεις πρέπει να συμμετάσχουν σύσσωμες. Έχουμε την υποψηφιότητα Αλσιζή για τις προεδρικές. Υπάρχουν άλλες υποψηφιότητες που θα μπορούσαν να προκύψουν από άλλες πολιτικές πηγές. Έπειτα μας είπατε ότι το πολιτικό τοπίο αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε φάση σύνθεσης με την ε, συμμετοχή των Ισλαμιστών. Ήθελα να μου πείτε. Πώς θα διαμορφωθεί αυτό το τοπίο μας ενδιαφέρει εν ώψη και των προεδρικών εκλογών. βέβαια το Σύνταγμα προβλέπει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και θα πρέπει να τηρηθεί. Πάντως, κύριε Μωράν, πιστεύω το πιο σημαντικό για να εξασφαλίσουμε την πρόοδο της διαδικασίας μετάβασης προς τη δημοκρατία είναι να εξασφαλίσουμε την οικονομική ανάκαμψη της Αιγύπτου. Γιατί είναι σημαντικό να σταματήσουν οι τρομοκρατικέ επιθέσει, να αποκατασταθεί μια ασφάλεια και η εμπιστοσύνη των πολιτών. Αυτό θα είναι η σημαντικότερη βάση για την ε, δημοκρατική μετάβαση. Σας ευχαριστώ πολύ για το έργο σας. Δυστυχώς βέβαια διαπιστώνουμε ότι οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία επισκίασαν ε, τη σημασία και τη, απόσπασαν την διεθνή προσοχή από τη Συρία και την Αίγυπτο και την έστρεψαν προς την Ουκρανία. Αλλά είναι σημαντικά τα γεγονότα και εξελίξεις στην ε, Αίγυπτο. Θα ήθελα να σας ευχαριστώ πάντως για την ενημέρωση αυτή στην Αίγυπτο δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική λύση. Μόνο το φιλοπορίας, η συνταγματική αναθεώρηση και οι επικείμενες ε, εκλογές. Σας ευχαριστώ και ευχαριστούμε για το έργο που επιτελείτε στην Αίγυπτο. Thank Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε, και σας ευχαριστώ που είσαστε εδώ πέρα και μας δίνετε μια αρκετά πλήρη επισκόπηση της σημερινής κατάστασης όπως την αντιμετωπίσετε εσείς. Η τελευταία μου επίσκεψη στην Αιγυπτό ήταν επίσης όταν η Task Force δημιουργήθηκε και έκτοτε προσπαθώ να παρακολουθώ τις ε, εκάστοτε εξελίξεις. Κάτι που μας ανησυχεί ιδιαίτερα, όχι μόνο εμένα, αλλά και πολλούς συναδέλφους, είναι η κατάσταση στο ΣΥΝΑ. Είπατε εν συντομία ότι επιδεινώνεται Νομίζω ότι ένα τμήμα του προβλήματος οφείλεται στις ε, περιορισμούς σε ό,τι αφορά την ασφάλεια λόγω των συμφωνιών μεταξύ του Ισραήλ και της Αιγύπτου. Αυτό εξακολουθεί να ισχύει ή μπορεί πλέον η Αιγυπτός να αποστέλει πιο πολλά στρατεύματα και πιο πολλές αστυνομικές δυνάμεις και το κράτη αυτό. Κάτι που ε, προκαλεί ανησυχία για το ΣΥΝΑ είναι η απάνθρωπη αντιμετώπιση των προσφύγων, κυρίως από το Σουδάν και από την Ερυθρέα, που προσπαθούν είτε να μεταβούν στο Ισραήλ είτε στην Αίγυπτο και που καταλήγουν όμοιροι των Βεδουίνων ως επιτοπλίστων, συμμοριών Βεδουίνων. Και αποδρούν ουσιαστικά με μεγάλη σκληρότητα και πλήρη τιμωρησία σχεδόν. Ρωτώ λοιπόν, αυτό ανησυχεί γενικά το κοινό και την κοινή γνώμη στην Αίγυπτο ή μήπως θα το πιάνει το ραντάρ της Αιγύπτου. Και πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την κατάσταση αυτή. Πώς μπορούμε να εκριζώσουμε τα φαινόμενα αυτά. Αυτή λοιπόν είναι μία ερώτηση που έχω να θέσω. Κάτι άλλο. Αναφέρεται σε ένα θέμα το οποίο θίξατε ακροθυγός. Η μεγάλη ευαισθησία που επικρατεί στην Αίγυπτο σε ό,τι αφορά οποιαδήποτε εξωτερική παρέμβαση και χρηματοδότηση δραστηριοτήτων και μη κυβερνητικών οργανώσεων. Έχει αλλάξει τίποτα. Έχει αλλάξει τίποτα. Έχει βελτιωθεί τίποτα σε ό,τι αφορά την κατάσταση των διεθνών μη κυβερνητικών οργανώσεων που εξακολουθούν, ελπίζουμε, να δραστηριοποιούνται στην Αίγυπτο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ. Ένα θερμό καλωσόρισμα, γιατί ήταν συναρπαστικό να ακούμε αυτή την σφαιρική παρουσίαση και αποτίμηση των όσων συμβαίνουν στην Αίγυπτο. Πρέπει να πω προσωπικώς, εγώ και η ομάδα μου, Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι με την σταθεροποίηση της ε, κατάστασης και με το νέο σύνταγμα. Κατά την άποψη των ε, Βρετανών ε, κοπτών από την Αίγυπτο στην εκλογική μου περιφέρεια, αυτό είναι ένα βήμα προόδου, αν και υπάρχουν και κάποιες ανησυχίες. Πάντως, ξέρουμε ότι σήμερα υπήρχε καταδίκη, δεκαετής κάθε, για δεκαετή κάθεξη και καταναγκαστικά έργα ε, κάποιων αστυνομικών που κατηγορήθηκαν για το θάνατο κάποιων από τους αδερφούς μουσουλμάνους. Δεν ξέρω λοιπόν αν ε, τέτοιου είδους ε, υποθέσεις δείχνουν πρόοδο από την πλευρά του κράτους δικαίου, όμως Πολλοί είναι αυτοί που ακόμη είναι φυλακισμένοι και θα πρέπει να δούμε με τι κατηγορίες θα δικαστούν και κατά πόσον. Έχω δύο ερωτήσεις τώρα για την οικονομία και τον τουρισμό. Τα πράγματα επανέρχονται στο κανονικό λόγο της σταθεροποίησης, διότι αυτό ήταν ένα καταστροφικό πλήγμα για την Αίγυπτο εδώ την διάρκεια της Επανάστασης. Αλλά η οικονομία πρέπει να σταθεροποιηθεί με ένα τόσο μεγάλο πληθυσμό. Ελπίζουμε ότι και η οικονομική άντιση μπορεί να φέρει σταθερότητα στη χώρα ούτως ή άλλως. Και επίσης, ποια είναι η τοποθέτηση της Αιγύπτου στην ε, περιοχή του, του αραβικού κόσμου και πώς βλέπει την ε, συνεργασία των χωρών του κόλπου με τη Σαουδική Αραβία, το Κουβέι, το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Ερμυράτα το Κατάρ φαίνεται να, συνδέ, να στηρίζει και πολύ συστηματικά την ε, μουσουλμανική αδελφότητα. Ενώ υπάρχει και υποστήριξη για μια νέα δημοκρατική κυβέρνηση. Πιστεύετε ότι το Κατάρ θα χρησιμοποιήσει τα, το βαθύ του πλούτο για να στηρίξει τις δικές του τις δραστηριότητες της MB κυρίως των, της των μουσουλμάνων ή θα πάρει κάποια άλλα θέση ως προς τη συνταγματική μεταρρύθμιση. Ευχαριστώ κύριε Σμιγιάν Μόν. Σας ευχαριστούμε κύριε Πρέσβε για την ανάλυση που μας κάνατε της κατάστασης ε, και τις ε, βραχυπρόθεσμες ε, προοπτικές. Πριν από τρία χρόνια όταν ξεκίνησε ε, η Αραβική Άνοιξη είδαμε πολλές διαφορές και πριν από 1,5 χρόνια είχαμε και την ίδρυση της, ε, το άνοιγμα της ε, αντιπροσωπείας μας και πολλών γραφείων. Θα ήρθε η ώρα όμως να κάνουμε ένα απολογισμό του ρόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα τελευταία τρία χρόνια στην Αίγυπτο. Γιατί παρά ε, την, ε, τις προσδοκίες μας από την Task Force ε, και τα 6 δισεκατομμύρια ευρώ που δώσαμε, νομίζω ότι δεν ε, είχαμε τις ε, αναμενόμενες εξελίξεις. Είδαμε το δρόμο που πήραν ο Μόρση και οι αδελφοί μουσουλμάνοι, δεν επηρεάσαμε ίσως αρκετά την κατάσταση ίσως ε, και λόγω της μεγαλύτερης παρουσίας των χωρών του Περσικού κόλπου. Και αυτό το μάντρα περισσότερο για περισσότερο, το more for more ε, μας εξυπηρέτησε και το θέμα της ε, έμφαση που δώσαμε στην παρουσία μας εκεί στη γειτονία εξυπηρέτησε κανένα σκόπο ή μήπως ήταν αποτυχία. Μήπως αυταπατώμαστε το περασμένο Φεβρουάριο, σε ένα ψήφισμά μας, στην πρώτη τελευταία παράγραφο, ζητούσαμε από την ε, κυρία Άστον να συνεχίσει τις διαμεσολαβητικές, τις διαμεσολαβητικές τις προσπάθειες για να επιλύσει την πολιτική κρίση. Υπάρχει δυνατότητα να έχουμε λόγο και να επηρεάσουμε τις εξελίξεις ελπίζουμε να μην επιβεβαιωθεί ένα καταστροφικό σενάριο και επανάληψη στην Αίγυπτο της κατάστασης της Αλγερίας πριν από 20 χρόνια. Βέβαια, δυστυχώ ε, επαναλαμβάνεται η ιστορία και ελπίζω να διαψευθώ. Θα ήθελα λοιπόν αυτό να μας πείτε. Μήπως επαναληφθεί η τραγική εμπειρία που είχαμε ε, για την Αλγερία τη δεκαετίας του 20. Ευχαριστώ. Κύριο κύριος Πρόεδρε, τι ευγενικό. Τρεις ερωτήσεις, αν με επιτρέπετε. Πρώτα απ' όλα, όταν ποτέ πηγαίνω στη λόγια της Γάζας, πρέπει να περάσω από την Αίγυπτο μέσω της Ράφα και από άλλα δύσκολα σημεία διόδου. Λόγω των προβλημάτων με τους αδερφούς μουσουλμάνους στην Αίγυπτο που ελέγχουν τις διόδους προς τη Γάζα, ήθελα να μου πείτε λίγα περισσότερα για τις επιπτώσεις, διότι η Αίγυπτος είναι το μόνο σημείο πρόσβασης, ή τουλάχιστον ήταν ως τώρα για να υπάρξει και οικονομική και οποιαδήποτε άλλη στήριξη προς τη Γάζα. Οι Ισραηλινοί απαγορεύουν την δίωδο και από αυτή την πλευρά, όπως ή άλλως. Και δεδομένων των εξελίξεων στην Αίγυπτο υπάρχει επίδραση και σε αυτό το τομέα. Υπάρχει κάτι να μου πείτε. Δεύτερον, ξέρω ότι είναι μια μικροσκοπική, μικροσκοπικότατη μειονότητα, αλλά οι εξτρεμιστές μουσουλμάνοι λένε ότι πρέπει να ανατινάξουν τις πυραμίδες γιατί είναι κάτι το απαράδεκτο. Ε, ούτως ή άλλως αρχαιολογικά μνημεία υπάρχουν σε όλη την ε, περιοχή της Μεσογείου, σε όλες τις ε, ακτές της δεν ήταν τέτοια η έκταση της καταστροφής ε, των αρχαίων μνημείων στην Αίγυπτο, όπως στη Λιβύη βεβαίως, αλλά είναι μια φανταστική περιοχή από ιστορικής άποψης. Τι μπορεί να γίνει γι' αυτό. Και τρίτον, μπορείτε να επεκταθείτε λιγάκι στα προβλήματα της υδροδότησης και του νερού, γιατί ο αρχικός στόχος των Αιγυπτίων ήταν ε, να γίνουν αυτάρκη στον τομέα αυτό, όμως τα προβλήματα ε, διαρκώς πολλαπλασιάζονται στον τομέα του νερού. Πιστεύετε ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτό ως μέσο πίεσης ε, με τον ένα τον άλλο τρόπο και μέσω των αποφάσεων που πρόκειται ενδεχομένως να εγκριθούν. Μπορείτε να μας πείτε λίγα περισσότερα γι' αυτό. Ευχαριστούμε. Κυρία Σάκη. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Κύριε Πρέσβη, σας ευχαριστούμε που είσαστε εδώ πέρα μαζί σας και σας ευχαριστούμε για την παρουσίαση που μας δίνετε. Επιβεβαιώνει λοιπόν τις ανησυχίες μας σε σχέση με αυτά που συμβαίνουν στην, Ευρω... στην ε, Αίγυπτο. Εγώ θα ήθελα να συμφωνήσω αρκετά με αυτά που είπε ο συνάδελφο Μιλαμόν και εγώ καλωσορίζω την πρόσκλησή σα για μεγαλύτερη συμμετοχή εδώ πέρα του Κοινοβουλίου για να έχουμε την ευκαιρία και να δούμε και την Ελλάδα άνστον να ε, έρθει εδώ στο Κοινοβούλιο για να μιλήσει για τις ανησυχίες μας, γιατί έχει περάσει πάρα πολλές χρόνος και είναι η πρώτη ευκαιρία που έχουμε να σχολιάσουμε τα σχόλια της Λαντιζάστον μετά το συνταγματική συνέλευση σε ό,τι αφορά τα σχόλια αυτά είναι περίεργα τουλάχιστον αναφέρει ότι παρακολουθήσαμε τα γεγονότα αυτά, τα περιστατικά αυτά από μια αποστολή παρατηρήση των εκλογών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συγχαίρουμε την ακολούθηση της διαδικασίας με σωστό τρόπο, δεν υπήρξαν οποιασδήποτε προβλήματα που να επηρεάζουν σημαντικά το αποτέλεσμα και φυσικά καταδικάζονται οι διαμαρτυρίες και τα γεγονότα τα βία περιστατικά που οδήγησαν σε θανάτους από όλες τις πλευρές. Και να αναφέρω ότι τα περιστατικά πριν από το δημοψήφισμα θα πρέπει να ερευνηθούν πιο πολύ από τις αρχές και σημειώνω ότι υπάρχει μεγάλη πλειοψηφία υπέρ το οποίο ε, σαφώς και υποστηρίζει το σχέδιο του συντάγματος, μετά επισέρχεται στην ουσία του θέματος. Αυτό που θεωρώ είναι απαραίτητο και περίεργο είναι το εξής. Αυτή είναι η αντιδρασή μας σε μια αποδοχή 90% ενός τέτοιου συντάγματος, όπου ξέρουμε ε, με βεβαιότητα ότι παρεμποδίστηκαν και παρακολούθηκαν ε, λύθηκαν οι αντίπαλοι το, του συντάγματος αυτού. Και αν δούμε τους ακτιβιστές με τους οποίους έχουμε επαφές τα τελευταία πέντε χρόνια και αν κοιτάξουμε και τα σχόλια υψηλόβαθμων αξιωματούχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δηλώνουν ότι η κατάσταση είναι χειρότερη παρά ποτέ και αυτό το κοιτάμε σε ένα περιβάλλον που δεν είναι έτσι κι αλλιώ ιδιαίτερα ρόδινο. Η κατάσταση είναι χειρότερη παραποτέ. Δεν ε, καταλαβαίνω με οποιοδήποτε τρόπο πόσο μεγάλο είναι το χάσμα μεταξύ των δηλώσεων αυτών και τη πραγματικότητα αυτή. Τι μήνυμα αποστέλουμε λοιπόν και με μεγαλύτερη έκπληξη μου προκάλεσε το γεγονός ότι δεν έγινε οποιοδήποτε σχόλιο και παρατηρήσει για τις συνταγματικές δηλώσεις του Μόρση. Τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να δώσει μεγαλύτερη ευελιξία με μεγαλύτερη φωνή, μεγαλύτερη ελευθερία έκφραση στον λαό των χωρών αυτών και θεωρώ ότι η έλλειψη πολιτικής ηγεσία και η έλλειψη σαφήνεια για το τι σημαίνει το more for more ενώ ουσιαστικά το υποστηρίζουν οι Ευρωπαίοι πολιτικοί σαν μια ενιαία λύση που ταιριάζει σε όλες τις χώρες της ε, γειτονία μας που αντιμετωπίζουν προβλήματα, σας παρακαλώ, για βοηθήστε με. Για πείτε μου, γιατί θα γίνουν πολλές εκλογές στο εγγύς μέλλον, κατά πάσα πιθανότητα πρώτα οι προεδρικές και μετά οι κοινοβουλευτικές, αντίθετα με όσα είχαν συμφωνηθεί και ελπίζω ότι το πλαίσιο στο οποίο θα λάβουν χώρα οι εκλογές αυτές θα ληφθεί πιο σοβαρά υπόψη προτού γίνουν δηλώσεις για το αποτέλεσμα και για τη συμμετοχή σε, ε, ότι, σε σχέση με τις δηλώσεις που έγιναν στις 19 Ιανουαρίου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για αυτή τη σειρά των τόσο τεκμηριωμένων και επίκαιρων ερωτήσεων. Δεν ξέρω αν θα μπορέσω να τις ε, απαντήσω όλες, αλλά θα δω τι θα κάνω. Κύριε Σαλαφράνκα, για το θέμα της επίσκεψης Λαμπρινίδη. Δεν ξέρω αν ο Σταύρο είχε την ευκαιρία να σα μιλήσει πρόσφατα. Ξέρω όμω ότι έχει επαφέ με όλου. σας. Νομίζω το καλύτερο θα ήταν να τα πει ο ίδιο. Έκανε μεγάλη προσπάθεια πάντως όταν ήρθε. Και είδαμε τον Υπουργό των Ιστορικών, τον Γενικό Εισαγγελέα να τον επισκέπτεται. Μιλάμε για δύο βασικού ε, παράγοντες όταν, σε ό,τι αφορά τι ε, φυλακίσεις. Και έκανε μεγάλη προσπάθεια να επισκεφτεί και κάποιου από του κρατουμένου, ώστε να απελευθερωθούν ενδεχομένω και έξι αυτοί κρατούμενοι. Τον στηρίζουμε. Και ελπίζουμε ότι θα γίνουν εφικτά όλα αυτά, διότι το Υπουργείο Εσωτερικών ε, έκανε μια, ένα δημοσίευμα στον τύπο, θα έδωσε ένα δημοσίευμα στον τύπο όταν έκανε την επίσκεψή του, λέγοντα ότι θα δοθούν διευκολύνσεις στους κρατουμένου. Προσπαθούμε λοιπόν να πιέσουμε μέσω διπλωματικών υπηρεσιών και πρέσβεων και κάνουμε ό,τι μπορούμε. Αυτό είναι κάτι επιπλέον σε σχέση με τι ιδέε που έχει για τι δεσμεύσει προ την νομοθεσία και το καθεξή. Σύμφωνα μαζί σα, το Σύνταγμα φαίνεται πολλά υποσχόμενο, ιδίω σε σχέση με το παρελθόν. Αλλά εκλογέ <coughs> και να έρθω στο θέμα των δηλώσεων τη 19 η Ιανουαρίου και το καθεξή. Η ψήφος, ψηφοφορία για το Σύνταγμα, όπω υπόθηκε, παρακολουθήθηκε από ειδικού περιεκλογών. Εμεί δεν μπορέσαμε βεβαίω να στείλουμε γέρο αποστολή, αλλά όλα αυτά βρίσκονται σε εξέλιξη. Δεν ξέρω αν η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση θα μπορέσει να σα δώσει περισσότερε λεπτομέρειε για αυτήν την αποστολή. Ήταν όμω μια περιορισμένη επίσκεψη με λίγου συμμετέχοντε χρήσιμη όμως που θα μας δώσει και κάποιες ενδεχομένως γνώσεις για το τι μπορούμε να κάνουμε στο μέλλον. Τώρα αν θα είναι συμμετοχικές και πολυφωνικές οι εκλογές ξέρουμε ότι υπάρχει για την ώρα ένας υποψήφιος, ο κύριος Εμπάχη, ίσως να υπάρξει και δεύτερος υποψήφιος, ίσως να προκύψουν και άλλοι, ίσως κάποιοι πιστεύουν ότι κάποιο υποψήφιο θα προκύψει προσπαθώντα να προσελκύσει και ε, το μουσουλμανικό κομμάτι του εκλογικού σώματο. Του Ισλαμιστέ. Όμω, ε, Ισλαμιστικά κόμματα υπάρχουν. Οι Σαλαφίτε επίση είναι μέρο τη όλη διαδικασία και άλλα κόμματα είναι ενεργά και μπορεί να έχουν συμμετοχή στι εκλογέ. Το κόμμα της ε, ελευθερίας, της δικαιοσύνης, είναι ένα κόμμα που μπορεί να προτείνει υποψήφιο για τις προεδρικές εκλογές, αν και δεν είναι τίποτε βέβαιο ακόμη. Για την κατάσταση στο ΣΥΝΑ Δεν το ανέφερα. Γνωρίζουμε πολύ καλά το ψήφισμα της 13ης Μαρτίου του Κοινοβουλίου για το θέμα της εμπορίας ανθρώπων και είναι κάτι που μας απασχολεί τρομερά και τα κρατημέλη και όλους μας. Είχαμε μια σειρά από συζητήσεις με το Υπουργείο Εξωτερικών Υποθέσεων και με άλλους ευθύνοντα για το θέμα αυτό, όμω η κατάσταση είναι φρικτά περίπλοκη στο ΣΥΝΑ. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η πρόσβαση. Πώ να πάει κανεί ε, στη θάλασσα και να δει τι γίνεται. Να δει, στην, ε, να δει τι συμβαίνει στην πράξη. Είναι και περίπλοκο και πολύ επικίνδυνο και για του διπλωμάτε, ε, και οι ομάδε που βρουν εκεί δεν είναι για αστείο. Δεν αστείευονται μάλλον. Ε, Είχαμε μακροσκελέστατες συζητήσει στην Αίγυπτο για το θέμα αυτό. Νομίζω το ψήφισμα είναι καλό. Καταδεικνύει τη σωστή κατεύθυνση και αυτή θα ακολουθήσουμε να επιδιώκουμε. Εάν η κατάσταση στο Σινά συνδέεται με το Camp David. Δεν νομίζω. Διότι η συνεργασία των δυνάμεων ασφαλεία Αιγύπτου-Ισραήλ είναι αρκετά αποτελεσματική για την ώρα. Νομίζω λοιπόν ότι σχετίζεται με πολλά άλλα στοιχεία η πρόσβαση στην Γάζα. Και υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που παίζουν ρόλο εδώ. Ε, ε, και οι Ευρωπαίοι μεταξύ άλλων. Και αυτό ε, περιπλέκει τα πράγματα στο Σινά. Επί μια δεκαετία το, αγνοή, το αγνοήθηκε η Χερσόνησο του Σινά. Και όμω τα πράγματα είναι πάρα, πάρα πολύ περίπλοκα. Οι Αιγυπτιακέ δυνάμει ασφαλεία κάνουν ό,τι μπορούν, αγωνίζονται, αλλά σε κάποιο βαθμό νομίζω ότι χρειάζονται και περισσότερη πείρα. Αυτό προσπαθούν να συγκεντρώσουν και τα πράγματα είναι επικίνδυνα, πολύ επικίνδυνα, η κατάσταση είναι έκρηθμη. Ε, η κατάσταση των ε, μη κυβερνητικών οργανώσεων ε, διεθνούς Τα πράγματα δεν είναι σταθερά. Για τον Υπουργό ε, Αλληλεγγύης και Εσωτερικών που ε, διορίστηκε την περασμένη εβδομάδα πρέπει να πω ότι θα δούμε πώς θα δικήσει αυτό το σημαντικότατο Υπουργείο, που αυτό είναι υπεύθυνο για τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Έχει αρκετή πείρα η υπουργό αυτή. Από την, άλλη αυτή. από την άλλη πλευρά, το Κοινωνικό και Αναπτυξιακό Ταμείο έχει κάνει μεγάλη πρόοδο συνεργαζόμενο με τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις τα τελευταία χρόνια. Πρόκειται πάντως για κάποια με πολύ προηγμένες απόψεις ό,τι αφορά τις διεθνείς, ε, διεθνείς με κυβερνητικές οργανώσεις. Θα δούμε λοιπόν πώς θα πάνε τα πράγματα και ποια δράση θα προτείνει για να προχωρήσουν τα πράγματα. Για την εκδόξη του κ. Τάνοκ. Είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα, πάρα πολύ σοβαρά. Παρακαλώ, πείτε στους φίλους σας να επισκεφθούν το Λούξο. Το 80% των ε, σκαφών είναι αυτή τη στιγμή προσαραγμένα μπροστά στο παλάτι. Είναι μια τραγωδία. Υπάρχει ένα παλιό αστείο στην ε, Αίγυπτο. Ότι χρειάζεται κανείς ε, πέντε, με ένα πεντά, πεντάλιρο ανεβαίνει σε καμήλα. Ε, αλλά για να κατέβει χρειάζονται 50 λίρες. Τώρα θα φτάσουμε τα 500 λίρες. Τα πράγματα πάνε πολύ δύσκολα, διότι στην Άνω Αίγυπτο τα πράγματα είναι ιδιαίτερα περίπλοκα και αυτή τη στιγμή και αλλού. Το Ασάν το ίδιο μετά τα πρόσφατα επεισόδια. Είναι τεράστιε λοιπόν οι δυσκολίε και το Υπουργείο Τουρισμού κάνει ό,τι μπορεί. Ο υπουργό είναι ε, ενεργότατο, είναι εντυπωσιακό, όπω και άλλοι προσπαθούν να κρατήσουν τα οχυρά του, αλλά είναι δύσκολα τα πράγματα και αυτό εξηγεί και την αύξηση τη φτώχεια που είδαμε τα τελευταία δύο χρόνια. Αντικατοπτρίζεται ε, το πώ 9 εκατομμύρια άνθρωποι που εξαρτώνται από τον τουρισμό έχουν πληγεί μιλάμε ότι είναι ο, μεγαλύτερος, ο δεύτερος μεγαλύτερος εργοδότης της χώρας μετά τη Γεωργία. Τεράστιο λοιπόν δυναμικό και τεράστια καταστροφή. Δεν θα επανέλθει ο τουρισμός και δεν έχει προφανώς επανέλθει, αλλά δεν θα επανέλθει αν δεν υπάρξει η ε, αποκατάσταση μιας ε, ελάχιστης ε, σφάλειας τουλάχιστον. Όπως και στη Χερσόνησο του Σίνα η Ερυθρά Θάλασσα είναι κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό. Και για, ε, για τα κράτη της συνεργασίας του κόλπου, το Κατάρ, ξέρουμε πως συνεχίζει να στηρίζει την, ε, τους, τους μουσουλμάνους. Είναι κάπως απομονωμένο βέβαια. Δεν ξέρω τι επίδραση θα έχουν, αλλά δεν θα ήθελα να κάνω εικασίες. Πάντως ε, τα πράγματα είναι σοβαρά εδώ. Οι Αιγύπτιοι έχουν αποπληρώσει ένα μεγάλο μέρος του χρέους, του δωρεάς που είχε δώσει το Κατάρ προς την ε, δημοσιαδικήση του. Ε, και κάποια από τα χρήματα δόθηκαν από άλλα κράτη του κόλπου για να αποπληρωθεί το Κατάρ. Η σχέση λοιπόν με το Κατάρ είναι ιδιαίτερα δυσχερή για του Αιγυπτίου αυτή τη στιγμή. Κύριε Μιλανών, σα ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την στρατηγικότατη ερώτηση που μου θέσατε. Τι ρόλο θα διαδραματίσουμε τα τελευταία χρόνια. Διαδραματίσαμε τα τελευταία χρόνια. Είμαι από το Φεβρουάριο του 2012 στην Αιγυπτοκιά. Για να είμαι απολύτω ειλικρινή, έχουμε κάνει ό,τι καλύτερο μπορούσαμε Χρησιμοποίησαμε τους καλύτερους αξιωματούχου μας. Ξέρετε τι προσπάθησε έκανε η Λεδιά στον πέρυσι για την συμφιλίωση και ξέρετε πώς επιμείναμε σε αυτό. Κάναμε ό,τι καλύτερο μπορέσαμε και ε, προσπαθήσαμε να προσελκύσουμε όλους προς αυτή την προσπάθεια. Ε, δεν πέτυχε βέβαια ε, για μια σειρά από λόγου. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε περισσότερα. Ίσως να έχετε διαφορετική άποψη, αλλά σε αυτό το μέτωπο δεν μπορούσαμε να κάνουμε περισσότερα. Γιατί γιατί αν τα πράγματα επανέλθουν και όλες οι πλευρές ζητήσουν το ίδιο πράγμα, μπορεί και να πετύχει. Ίσως την επόμενη φορά μπορεί να τα καταφέρναμε, αλλά αναφέρεται και την Αλγερία και είναι πολύ διαφορετικά αυτά που έγιναν στην Αλγερία ή στην Αίγυπτο. Στην Αίγυπτο οι αδελφοί μουσουλμάνοι ήταν μια δύναμη μεταξύ των πολιτών, δεν ήταν αναγκαστικά ένοπλοι ήταν ε, κυβέρνηση για έναν ολόκληρο χρόνο. Οπότε τα πράγματα είναι αρκετά διαφορετικά από ότι στην Αλγερία. Έχουμε πάρα πάρα πολλά να μάθουμε ακόμη όλοι μας και σε αυτό το μέρος του κόσμου και θα νομίζω θα σταματήσω εδώ. Σερ Ρόμπερτ για τη Γάζα δεν θα απλουστευτούν τα πράγματα. Οι ενέργειε τη ε, Χαμά και η παρουσία τη Χαμά απαγορεύτηκε στην Αίγυπτο. Βεβαίω, περιέργω, ε, στην ανακοχή που ήταν δικημένο διαπραγματεύσεων την περασμένη εβδομάδα πήραν μέρο και οι Αιγύπτιοι. Φαίνεται λοιπόν να υπάρχει ενδιαφέρον για, την, ε, για το σταθμό του ΑΚΑ, αλλά οι εσωτερικέ εξελίξει στην Αίγυπτο μπορεί να επηρεάσουν την κατάσταση. Μετά τι εκλογέ θα δούμε τι θα γίνει εάν θα έχουν ενεργότερο ρόλο και αν θα βελτιωθεί η κατάσταση σε αυτή την περίπλοκη σχέση. Για τα αρχαιολογικά μνημεία. Για πρώτη φορά έχουμε μια δυνατότητα αδερφοποίησης με, ε, με το Υπουργείο Αρχαιοτήτων. Θα σας τηρώ ενήμερο. Για τα νερά του Νείλου. Ένα πολύ περίπλοκο ζήτημα. Οι Αιγύπτιοι αισθάνονται ότι απειλούνται Διότι προφανώ το 95% του πόσου νερού τη χώρα προέρχεται από τον ήλιο, κάτι που δεν σα εκπλήσει. Οι προσπάθειε συνεργασία που θα δώσουν ωφέλη και στι δύο πλευρέ είναι κάτι που δεν αποδίδει. Οι, Αιθιο... από τη δική του πλευρά δεν φαίνεται να είναι ανοιχτοί στο να υπάρξει περισσότερη συνεργασία και δεσμεύσει με του Αιγυπτίου. Θα καθυστερήσει η οικοδόμηση φράγματο και η δικαιολογία είναι ότι είναι δικό τους ε, κυρίαρχο δικαίωμα να το οικοδομήσουν ή όχι, όμως θα πρέπει και πάλι να καθίσουν σε ένα τραπέζι και να συζητήσουν, να περάσουν σε ένα πλαίσιο συνεργασίας οι δύο πλευρές και πάλι δεν θέλω να υπερβάλλω και να το χρησιμοποιήσω αυτό ως δικαιολογία, αλλά ίσως μετά τις εκλογές να πρέπει να περιμένουμε και να δούμε αν είναι απλούστερο για την Αίγυπτο να προχωρήσει αυτή την κατεύθυνση. Προς τη στιγμή πάντως έχει πρόβλημα. Και πρέπει να παρακολουθούμε πάρα πολύ, πολύ στενά το θέμα αυτό θα ήταν ε, πρόβλημα εάν, υπήρχε πρόβλημα, αν κάτι προέκυπτε με το φράγμα. Δεν ξέρω αν θα έρθει η Λέδη στον ε, κυρία Σάκια, αλλά το μήνυμα πέρασε και θα τη το μεταφέρουμε. Η απόκριση στο δημοψήφισμα. Ναι, ήταν ε, μεγάλο το ποσοστό και είναι σαφές, αλλά υπήρξε και μοικοτάρισμα, μην το ξεχνάτε αυτό. Μεγάλος αριθμός πολιτών απλώς δεν ψήφισαν και δεν ήθελαν να ψηφίσουν. Αυτό λοιπόν είναι κάτι που δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Από την άλλη, νομίζω στη δήλωση δώσαμε και κάποια απόχρωση σε αυτά που είπαμε, στα λόγια μας συγκεκριμένα, ε, με κάποιους χαρακτηρισμούς. Νομίζω σημαντικό είναι να δούμε την ουσία. Τι σύνταγμα ψηφίστηκε τελικά, όπως είπα προηγουμένως. Ναι, υπήρχαν προβλήματα, αλλά υπάρχουν τομεί όπου πραγματικά είναι πολλά υποσχόμενα το Σύνταγμα, ιδίω για τι θεμελίδε ελευθερία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό πρέπει να το παρακολουθούμε πάρα πολύ στενά. Οι Αιγύπτιοι το ψήφισαν αυτό. Τώρα λοιπόν οι πολιτικοί φορεί, οι πολιτικοί θύνοντε πρέπει να δώσουν αποτελέσματα να πετύχουν αποτελέσματα. Και επανέρχομαι στο αρχικό μου σχόλιο, σε ό,τι αφορά το κοινοβούλιο, αυτό το κοινοβούλιο. Πρέπει να γίνουν μεγάλε προσπάθειε και συνεργασία με την Ηγετική Βουλή, ώστε να γίνουν και κάποιε χειροπιαστέ ενέργειε στην ε, χώρα. Νομίζω ότι το Σύνταγμα αυτό μα δίνει πραγματικέ ευκαιρίε να έχουμε πραγματική συνεργασία, αλλά δεν θέλω να υπερβάλλω. Και τώρα για το για το more for more, για την αρχή αυτή. Είναι σαφές ότι αν έχει κανεί μια τέτοια αρχή κατά νου, θα πρέπει να υπάρχει συνένεση, να υπάρχει ευφύς ε, εφαρμογή. Όχι με τρόπο ε, πιεστικό, με καταπίεση, αλλά να γίνει δεκτό και από την Αίγυπτο. Σίγουρα τα κονδυλιά μας είναι σημαντικά, σίγουρα η ποιότητα της βοήθειάς μας είναι υψηλή, ίσως υψηλότερη, όμως το ποσό έχει περικοπεί πάρα πολύ. 17 δις ε, δολάρια ήρθαν από τα κράτη του κόλπου την περασμένη φορά ο και έρχεται και άλλο ποσό. Δεν είναι όλα δωρεέ, αλλά κάποια φορά από αυτά είναι παραχωρητικά δάνεια. Ε, οπότε, σε ό,τι αφορά τα κονδύλια και την μόχλωση, ναι, είναι κάτι που μπορούμε να το έχουμε κατά νου. Τώρα, σε κάποιους πολύ συγκεκριμένου, ε, εντοπισμένου κιόλα τομεί, θα μπορούσαμε να τα είχαμε πάει καλύτερα αν ήμασταν πιο ευφυεί και είχαμε καλύτερη στόχευση των όσων θέλαμε να πετύχουμε. Ευχαριστώ. Ε, σας ευχαριστούμε κύριε Μωράν, κύριε Πρέσβε. Πριν να ε, κηρύξω το πέρας της πρωινής συνεδρίασης, να σας υπενθυμίσω ότι στις 3 θα ξεκινήσουμε ε, στις 3 με παρουσία του κύριου Φιένερ του Διαχειριστικού Διευθυντή της ΕΙΕΔ. Καλώς μεσημέρι.